Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας, την Δήμερη. Σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και όσον αφορά την διερμηνία, προτεραιότητα δίνεται πάντα στα πλήρη μέλη της Επιτροπής μας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα. Τη απουσία παρατηρήσεων θεωρώ την ημερήσια διάταξη εγκεκριμένη. Η γραμματεία έχει μοιράσει και τα πρακτικά της προηγούμενης ε, συνεδρίασής μας της 14 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας ή τις επιφυλάξεις σας μέχρι το τέλος της αυριανής μας συνεδρίασης, αύριο το μεσημέρι δηλαδή. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στο διευρυμένο Προεδρείο που θα έχουμε θα ήθελα να συζητήσουμε πρόταση του κυρίου Γκάλερ να συμπεριλάβουμε συζητήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΠΕΣΚΟ. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα που προτείνω. Είτε να μπει ένα χωριστό σημείο χρηματοδότηση της ΠΕΣΚΟ ή προτιμότερο νομίζω ακόμα να υποβάλουμε προφορική ερώτηση ως ΣΕΝΤΕ προκειμένου να συζητηθεί αυτή κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Οπότε, πρώτα απ' όλα, αν συμφωνεί ο κύριος Γκάλερ, νομίζω ότι θα ήταν μια καλή λύση αυτή. Στο δίλημά σας, κύριε Γκάλερ. Αλλά θα συζητηθεί, όπως είπα, στο διευρυμένο Προεδρείο μας σήμερα το βράδυ. συγγνώμη ε, για τη φωνή μου, θα κάνω κάποιες διακοπές. Να ξέρετε ότι έρχομαι από γρήπη και είναι η πρώτη μου μέρα στη δουλειά και πάλι. Ωραία, λοιπόν. Περνάμε τώρα στο πρώτο ουσιώδες σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της ΕΝΤΕ στο Ταλίν της Εστονίας και στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Στην Εστονία δεν πήγαμε μόνο στο Ταλίν, πήγαμε και στο Αμαρί. που είναι μια αεροπορική βάση. Και μπορέσαμε εκεί να επισκεφτούμε και αυτά τα μέρη. Συμμετείχαν εγώ ίδια, αλλά επίσης ο κύριος Γκάλλαρ, ο κύριος Τουνεκέλαμ, ο κύριος Χρουνζουλίκα, ο κύριος Σίντρικ Ταράντ, και ήμασταν τρεις μέρες στην αποστολή αυτή. Αρχίσαμε με το Ταλίν, με ανταλλαγή απόψεων με διάφορους υπουργούς της Εστονίας, με πολύ έμπειρους Εστονούς διπλωμάτες και είχαμε εξαιρετική παρουσίαση για τις διάφορες ε, πτυχές που έχουν να κάνουν με τις θέσεις της ε, Εστονίας απέναντι σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Και είχαμε και μια επισκόπηση όσον αφορά την κατάσταση ε, για την ασφάλεια. Στη συνέχεια πήγαμε στην αεροπορική βάση του Άμαρη, όπου εκεί συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της Ιταλικής Μοίρας που είναι εκεί και συναντηθήκαμε και με την Αμερικανική Μοίρα. μπορέσαμε έτσι να δούμε στρατιωτικά αεροπλάνα και Eurofighters και F-16 τα οποία βρίσκονταν στην αεροπορική αυτή βάση και ακούσαμε και ενημερωτικές παρουσιάσεις από τους εστονούς οι οποίοι δουλεύουν εκεί. Την επόμενη μέρα είχαμε ενημέρωση στο Υπουργείο Άμυνας. Ε, συναντηθήκαμε με υψηλά στάμενους ε, εμπειρογνώμονες, συμβούλους, αξιωματούχους και επισκεφθήκαμε κάτι που ήταν το πιο σημαντικό νομίζω στην ημερήσια μας διάταξη και ο στόχος της επίσκεψής μας εκεί. Πήγαμε σε ένα κέντρο αριστείας όσον αφορά την κυβερνόμηνα Και εκεί ακούσαμε νους αλλά και άλλους ειδικού στον τομέα αυτό. Θυμίζω ότι το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε αμέσως μετά την κρίση του 2007 και τις σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις που έγιναν τότε στις υποδομές της Εστονίας. Έκτοτε η χώρα αυτή, η Εστονία δηλαδή, βρίσκεται στην πρώτη θέση προκειμένου να εκπονήσει προγράμματα κυβερνόμενας και άλλα προγράμματα για να αντιμετωπίσει τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε με εκπροσώπους ε, της Επιτροπής Άμυνας του Κοινοβουλίου της Εστονίας. Ήταν πολύ παρόλο που η μέρα της επίσκεψής μας ήταν και ετήσια ημέρα για πέτειο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την εξωτερική πολιτική της Εστονίας. Υπήρχε σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο της χώρας. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες στην Εστονία για την υποδοχή τους και την θερμή τους φιλοξενία στο Ταλίν. Επόμενο θέμα στην εμερήσια διάταξη ήταν η επίσκεψή μας το, σε εκπροσώπους του κλάδου της άμυνας και συζητήσαμε μαζί τους για τις προοπτικές της Εσθονίας όσον αφορά την βιομηχανία άμυνας. πώς εντάσσονται στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ΠΕΣΚΟ. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Λισίνκι να το φέρει. Και εκεί είχαμε εκτενείς παρουσιάσεις στο Υπουργείο Άμυνας από το προσωπικό, από τον επικεφαλής την Άμυνα. Συναντηθήκαμε με την Επιτροπή Άμυνας του Φιλανδικού Κοινοβουλίου. Και επίσης επισκεφθήκαμε και συζητήσαμε εκτενώς, είχαμε ανταλλαγή απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας σχετικά με την κύβερνόμηνα. Ακούσαμε για τις εργασίες τους, τι έχουν ήδη κάνει και ποια τα σχέδιά τους για το μέλλον. Η πρώτη μας μέρα στο Ελσίνκι έκλεισε με συνάντηση με την ε, Ένωση που έχει να κάνει με την βιομηχανία άμυνας. Εκεί ακούσαμε λεπτομερώς για τις προτεραιότητες της φιλανδικής βιομηχανίας άμυνας. Και την επόμενη μέρα, την τελευταία της επίσκεψής μας, την αφιερώσαμε σε ανταλλαγή απόψεων με τον Φιλανδό επικεφαλής άμυνας. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να, συμμετάσχουμε σε συνάντηση όπως είχαμε προβλέψει αρχικά με την Αμυντική Ακαδημία. Και αυτό γιατί άλλαξαν τα σχέδια. όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην αποστολή έπρεπε κάποιοι να πάρουν το αεροπλάνα τους, οπότε δεν προλάβαμε. Αυτά όσον αφορά την ενημέρωση αυτή. Συνεπώς τώρα συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Κέλα μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ήμουν ευτυχής ε, να πάω στην Αστονία ε, και στη Φιλανδία υπό την ηγεσία σας. Για μας αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν ακριβώς η σύγκριση ανάμεσα στην Αστονία και στη Φιλανδία. Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που μας ήρθε από το Υπουργείο Άμυνας της Εστονίας, για παράδειγμα, για την ε, επίθεση στον κυβερνοχώρο πριν από μερικά χρόνια, του οδήγησε σε μια συγκεκριμένη πορεία. Τώρα βέβαια η Ρωσία επιτίθεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι κάτι κοινό μεταξύ όλων μας η υπόθεση αυτή. Όσον αφορά την αεροπορική βάση στο Όμαρη, και αυτή η εξέλιξη πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. είδαμε την Αμερικανική μοίρα που μόλις είχε φτάσει, που τρεις φορές το χρόνο πάει στο Άμαρι, τρεις-τέσσερις εβδομάδες κάθε φορά η παρουσία αυτή της αποτρεπτικής δύναμης του ΝΑΤΟ νομίζω ότι είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Όπως είπε και ο υπουργό Άμυνα, σε περίπτωση επίθεσης ε, χρειάζεται ενίσχυση. Και το θέμα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ενίσχυση. Στη συνέχεια, όσον αφορά τις αμυντικές δυνάμεις της Φιλανδίας. Η δικιά μου εντύπωση ήταν ε, ιδιαίτερα θετική, κάτι που δεν περίμενα. Γιατί όλοι καταλήξαμε στο ότι η Φιλανδία τελικά είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη όσον αφορά τις απαιτήσει του ΝΑΤΟ από άλλες χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Υπάρχει εθνική ενότητα όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, την εδαφική άμυνα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επ' αυτού δεν θα έχει κανείς που θα προσπαθήσει επίθεση δυνατότητες να πετύχει στη Φιλανδία. Εξυγχρονίζουν επίσης τον αμυντικό τους εξοπλισμό με έναν ε, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο εξοπλισμός έχει 600, το πυροβολικό 600 κομμάτια. 1600. Και η Φιλανδία είναι πάρα πολύ θετική απέναντι στην ΠΕΣΚΟ. Ακόμα και ανεξάρτητα από τον ΝΑΤΟ. Και είναι υπέρ της ε, συνεργασίας των βόρειων χωρών. Δεν βάζουν λοιπόν όρια και περιορισμούς στη συνεργασία με άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αναφερθήκατε στο κέντρο αριστείας για την ε, αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων ε, και για τις υβριδικές απειλές. Ε, ξεκίνησε τον Οκτώβριο που μας πέρασε, είναι πολύ νέο. Και είναι κάτι που γεφυρώνει τον ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και να μπορούν και να τις αναλύουν καλύτερα. Πώς δηλαδή αυτές οι υβριδικές απειλές λειτουργούν τελικά. Για παράδειγμα, είχαν ένα σεμινάριο στο Βίλνιους τον Νοέμβριο όσον αφορά τη ρωσική επιρροή στην περιοχή. Και με εξέπληξε όταν συναντήθηκα με την αμυντική βιομηχανία και τους εκπροσώπους της, γιατί διαπιστώσα ότι είναι πάρα πολύ δυναμική και πολύ καλά προετοιμασμένη. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι από τα κέρδη τους επενδύουν 15% στην έρευνα και την ανάπτυξη, που είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, αν το συγκρίνουμε με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που το καλύπτουν για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη φιλανδική βιομηχανία. Είναι πολύ θαρρυντικό το παράδειγμα αυτό δηλαδή. Πώς μια σχετικά μικρή χώρα μπορεί να προετοιμάσει καλά την άμυνά της. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, σίγουρα όλοι συμμεριζόμαστε τις δικές σας εκτιμήσεις. Πράγματι, ήταν ε, εξαιρετική η συνάντηση αυτή. Όλες οι επαφές μας ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες. Κλέρ Μούντι, τώρα η αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ. Σύντομο. Σύντομα. Και τα δύο αυτά κέντρα για την κυβερνοασφάλεια και για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών συνεργάζονται πολύ στενά ε, σε τομείς που μας ενδιαφέρουν πολύ εμάς. Αυτά που είδατε από την επίσκεψη των δύο κέντρων θα πρέπει να μας ευνεύσουν για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή δράση σε αυτούς τους τομείς. Ειδικά στην κυβερνοάμυνα. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά και οι υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Κύριο Στατίνα, αντιπρόεδρος. Πρόεδρε. Θα μιλήσω τσέχικα, παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Ο κύριος Κέρλαμ ανέφερε την ενότητα. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να πούμε ότι τα βαλτικά κράτη, ούτε καν η Εστονία, ε, μπορούν να τα καταφέρουν από μόνα τους. Αναφέρατε αυτή την ε, σημαντική στρατιωτική βάση, ε, αεροπορική στρατιωτική βάση της Εστονίας, ξέχασα το όνομα, μάλιστα. Και αυτό είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η αμοιβαία στήριξη, η αμοιβαία αρρωγή. Παλιά ε, τσεχικά αεροσκάφη χρησιμοποιούσαν αυτή την αεροπορική βάση. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούσαμε να δούμε διαγράμματα που αποδείκνυαν ότι τη στιγμή που το τσεχικό αεροσκάφος ε, έμπαινε στην Εστονία, φαινόταν ότι τα, τα ρωσικά ε, αεροσκάφη ε, σταματούσαν τις επιδρομές τους ε, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Μειωνόταν τέλος πάντων πάρα πολύ η συχνότητα του φαινομένου αυτού των επιδρομών των ε, ρωσικών αεροσκαφών. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Thank you. Ευχαριστώ. Η Τούλα μπορεί να κάνει και αυτή ερωτήσεις ή να σκεφτεί και αυτή τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Η δική μου εντύπωση και για τα δύο κέντρα διαφέρει σχετικά. introduced. Η... η μεγάλη δουλειά που έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Ελσίνκι ήταν, είχε σαν σκοπό να δημιουργήσει κάποιες διαδικασίες για να υπάρχει μια πλησιέστερη σχέση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν και, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για τον επιμερισμό καλών πρακτικών με διάφορα κράτη-μέλη. τόσο ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ξεπεράσουν την απροθυμία που έχουν, την φυσική απροθυμία που έχουν στο να μοιράζονται τις πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Τώρα για το κέντρο, το εστονικό στο Τάλιν. Υπάρχει... Έχουμε εμπειρία από παλιά με αυτό το κέντρο. με εστίαση σε πρακτικά ε, project για την αντιμετώπιση των ε, κυβερνοπυλών. Για τη βάση στο Άμαρι, έχει έναν ισχυμένο ρόλο, ο οποίος ξεκίνησε μετά την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Εστονία. Προέδρου τότε και υποσχέθηκε ότι το Άμαρι θα γίνει μια βάση εκπαίδευσης για τα αμερικανικά στρατεύματα. Και οι περιπολίες και η αερονομία, οι επιχειρήσεις αερονομίας είναι πολύ σημαντικές υπήρχαν περιστατικά προβλήματα, ας πούμε, που είχαν δημιουργηθεί. Και, και εσείς, κύριε Στετίνα, επίσης έχετε δίκιο ότι η παρουσία άλλων χωρών στην Εσθονία και η επίδειξη αλληλεγγύης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει όμως, να υπάρχουν επιχειρήσεις αερονομίας και να μπορούν σε περίπτωση που έχουμε βία επεισόδια και παραβιάσεις ας πούμε του εναέριου χώρου να παρεμβαίνουν τα αεροσκάφη μας. Δεν κατάλαβα την πρώτη σας ερώτηση, πρέπει να ομολογήσω. είχε να, να κάνει με το κατά πόσο έχουμε, είμαστε αποτελεσματικοί στο να υπερασπιστούμε τις βαλτικές χώρες. Οι ίδιες οι βαλτικές χώρες ε, προσπαθούν να αυξήσουν τις δυνατότητές τους, τις στρατιωτικές δυνατότητές τους. Έχουν αποφασίσει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Για την Εστονία δεν είναι απαραίτητο παρότι είχε αποφασίσει η χώρα να το κάνει. Η Εστονία είναι μία από τις λίγες χώρες που φτάνουν τους στόχους του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν επίσης και πολλά στρατεύματα από τρίτες χώρες στις βαλτικές χώρες, στη Λιθουανία, στη Η Γερμανία επίσης στην Εστονία, είναι παρούσα στην Εστονία. Υπάρχει βάση ΤΑΠΑ, υπάρχει και βρετανική παρουσία εκεί, παρουσία βρετανικών στρατευμάτων δηλαδή στο, στην ΤΑΠΑ. Και εμείς θα θέλαμε να επισκεφτούμε αυτή την ε, βάση. Αυτό που έλειπε από αυτή την επίσκεψη, κατά τη γνώμη μου, ήταν η συμμετοχή και οι συζητήσεις στη βάση ΤΑΠΑ. Ίσως θα την επισκεφτούμε αργότερα. Σκεφτείτε το κύριε μου αυτό το θέμα. Και σας δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Νομίζω και στις δύο βάσεις και στα δύο κέντρα, το ένα για την αντιμετώπιση των υβριδικών πόλεμων και το άλλο για το κυβερνοχώρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαβίβαση των πληροφοριών. Είναι το θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών είναι πάρα πολύ απρόθυμες να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλους. Και τα δύο αυτά κέντρα όμως ε, λειτουργούν εθελοντικά το Κέντρο Αντιμετώπιση βρυδικών Απειλών στο Ελσίνκι αυτή τη στιγμή έχει 13 συμμετέχοντες με αύξουσα τάση. Είναι οι χώρες της Βαλτικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένε Πολιτείε και τα δύο κέντρα, μάλλον και οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει και στο κέντρο του Ταλίν που φτάνει τα 30 άτομα. Οι συνομιλίες είναι με βάση το Chatham House και πώς να το πω γίνεται και μια συζήτηση για το πώς ερμηνεύουμε τη δήλωση του Συμβουλίου που ανάγεται σε μια ε, τετραετία ότι ε, κατά περίπτωση οι επιθέσεις του κυβερνοχώρου και οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να εμπίπτουν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Και σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις είναι ένα μόνο τμήμα ενός πιο περίπλοκου συστήματος επίθεσης. Κάτι άλλο που είχε ενδιαφέρον στο κέντρο κυβερνοχώρου στο Ταλίν είναι ότι παίζουν εκεί κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δηλαδή. Κάνουν ασκήσεις υποτιθέμενες ε, κυβερνοαπειλής και επίθεσης εναντίον ενός ε, στόχου και υπάρχει μια ομάδα επιτιθέμενη, μια αμυνόμενη, κόκκινη, μπλε και μια ουδέτερη. Είναι καλή άσκηση αυτή και καλή πρόβα για το πώς ε, θα πρέπει κανείς να αντιδρά σε περίπτωση σοβαρών επιθέσεων. Εξεπλάγει και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από αυτό. Στο Ελσίνκι, για μένα, το σημαντικότερο ήταν ότι εμείς εδώ συζητούμε πάρα πολύ θεωρητικά για τις επιθέσεις κυβερνοχώρου. Και τι σημαίνουν αυτές. Ενώ εκείνοι έχουν ξεκαθαρίσει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Υπάρχουν διάφορες φάσεις και στάδια. Ποια είναι η πρώτη φάση. Η πρώτη φάση είναι να αυξήσεις ε, τον, ε, το ευάλωτο χαρακτήρα του αντιπάλου, να τον αποδυναμώσει στην εσωτερική συνοχή, την κοινωνική συνοχή, να δημιουργήσει κοινωνικές ταραχές κτλ. στο διαδίκτυο. Σε δεύτερη φάση ε, έχουμε χρήση βίας από στρατιωτικές ομάδες, οι παραστρατιωτικές, όχι τον τακτικό στρατό, με δολοφονίες, ενδεχομένως και ζημίες και καταστροφή κρίσιμων υποδομών κτλ. Αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες να είναι προετοιμασμένοι για τις συγκεκριμένες αυτές καταστάσεις και πώς αναπτύσσουν αυτά τα σενάρια για να λειτουργήσουν στην πράξη. Θα το δούμε ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα με τις πρακτικές ε, περιπτώσεις ε, και τις συγκεκριμένες. Πάντως ε, αυτή η πρωτοβουλία υπόσχεται πολλά. και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τον Οκτώβριο όταν ε, στα εγγένεια αυτού του κέντρου παρουσία της κυρίας Μογκερίνη, η κυρία Μογκερίνη εγγενίασε και παρουσία του Φιλανδού Προέδρου, όλα αυτά ξεκίνησαν ε, σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι πολύ ελπιδοφόρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κλείσουμε την ενημέρωση της για την αποστολή μας ε, στην Εστονία και την Φιλανδία. This, ε, Αυτό έγινε πολύ σύντομα ενημέρωση, πολύ σύντομα μετά την επίσκεψη και ήταν καλό αυτό. Και σας ευχαριστώ. Τώρα, Έχουμε το συντάκτη νομοδότησης για τη δημιουργία ενός πλαισίου ε, για τον έλεγχο των ε, ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο κύριος Βανόρδεν, ο συντάκτης της νομοδότησης και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. 12 εγκρίθηκαν εξ όσων γνωρίζω Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Βανόρντεν τι έχει να μας πει. Να μας παρουσιάσει την ε, γνωμοδότησή του και να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό προφανώς και οι συνάδελφοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Uh, Πάνω από 200 ε, τροπολογίες υπευλήθησαν οι προτάσεις για τροπολογίες Βέβαια, την περασμένη εβδομάδα μόλις πήραμε τις τροπολογίες και υπάρχουν πολλές και σε πολλές γλώσσες. Ακόμα δεν λάβαμε τη μετάφραση στα αγγλικά όλων των τροπολογιών. Και μαθαίνω ότι 1η Μαρτίου θα φτάσουν οι μεταφράσεις, που δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ από πλευράς χρονοδιαγράμματος αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Προφανώς μελέτησα ε, τις τροπολογίες και όπως πάντα υπάρχουν κάποιες τροπολογίες με τις οποίες μπορώ να συμφωνήσω, μπορώ να τις δεχτώ και βοηθούν γενικά. Κάποιες άλλες δεν βοηθούν πάρα πολύ. Ελπίζω όμως στα πλαίσια των συμβιβασμών πρώτα να μειώσουμε τον αριθμό των τροπολογιών που θα κληθούμε να ψηφίσουμε και να βρούμε και μια διατύπωση που μπορούν όλοι να τη δεχθούν. Θα συνεδριάσουν αύριο οι σκιώδες συγγητές στις 3.30 το απόγευμα και μέχρι τότε θα σας έχουμε κάνει προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες και θα τις ε, διανύμουμε. Ζητώ όμως την επίκαια σας γιατί είναι πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα και θα προσπαθήσω να ε, σας ε, τα στείλω μέχρι αύριο το μεσημέρι το αργότερο για να έχετε χρόνο να τις κοιτάξετε πριν συνεδριάσουμε στις 3.30 αύριο και οδησηγητές. Η Επιτροπή θα ψηφίσει την αναθεωρημένη γνωμοδότηση την εβδομάδα που αρχίζει ε, στις 19 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασής της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Ίντα και η συγητής ο κύριος Φρανκ Προύστ. Και ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, θα εγκριθεί το Μάρτιο, στις 19 ή στις 20, ε, θα τα συνεδριάσουν εκεί. Θα δώσω το λόγο πρώτα στους και όδης η κυρία Αντρική είναι πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τζέφρι Βανόρδεν για το σχέδιο γνωμοδότησης που σήμερα συζητούμε. Κάποια γενικά σχόλια για το θέμα αυτό. Η νέα πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη και αποτελεί καλή αρχή. Ωστόσο δεν πρόκειται να αποδειχθεί επαρκής για να αντισταθμίσει την αποκεντρωμένη και κατακαιρματισμένη προσπάθεια ε, ξένων δυνάμεων. Γίνονται κάποιες καλές προτάσεις, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο φιλόδοξη, ε, ούτε είναι ε, αυτός καθ' αυτός μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ανταλλάσσουν προφορίες και μόνο τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και προς το παρόν δεν γνωρίζουν τον πλήρη βαθμό ε, ούτε το μέγεθος της, ε, των άμεσων ξένων επενδύσεων και στρατηγικών επενδύσεων. Έχουμε εμεί ενδείξεις ότι οι εταιρείε που συνδέονται με την Κίνα ε, στρατηγικά επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, όχι μόνο στο πολιτικό τομέα, αλλά και στο στρατιωτικό. Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί έχουν τεχνολογία που βρίσκεται ήδη σε αεροσκάφη, σκάφη και υποβρύχια κινέζικα. Επίση, οι άμεσες ξένες επενδύσει αφορούν κρίσιμα λιμάνια, ε, όπω είναι ο Πειραιά ε, και το, το Ζέμπροχε στη Βέλγιο, ε, εργοστάσια που φτιάχνουν ρομπότ όπως το Όμιλος Κούκα στη Γερμανία, έχουν πολλές μετοχές και κρίσιμες από τις Deutsche Bank και αλλού και στο Ηνωμένο Βασίλειο το Skyscan και αυξάνεται και με ανησυχεί αυτή η τάση. Κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει ε, την τεχνολογική αιχμή στην οποία βρίσκεται και την ηγεσία. Και επιπλέον ο μηχανισμό ελέγχου άμεσων ξανεπενδύσεων είναι ένα θέμα ασφαλεία που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι είναι και θέμα εμπιστοσύνη. Υπάρχει θέμα ε, απορρίτου ε, των ε, πληροφοριών που ε, μοιραζόμαστε και θα πρέπει αυτό να προστατεύεται και να προβλέπονται και μέτρα πειθαρχικά. Επίσης, οι επενδυτές παρακάμπτουν συγκεκριμένα κράτη και βρίσκουν μια χώρα που είναι πιο ευάλωτη για να διεισδύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούν αυτά τα παραθυράκια και πηγαίνουν σε ε, πιο ευάλωτους κλάδους της οικονομίας και της βιομηχανίας που δεν καλύπτεται από τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Σήμερα ε, μπορεί να μην φαίνεται ο αντίκτυπο, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει ίσου κανόνου παιχνιδιού, θα πρέπει να προχωρήσει πολύ πέρα από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ρυθμίζει τα θέματα του βασικού μετόχου, την πρόσβαση στις ε, βιομηχανίες ε, και χρειάζεται ένας πιο ισχυρό μηχανισμός και μεγαλύτερη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλο ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βγάλει τα διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες. Βλέπε Gazprom και πώς ε, υπάρχει αυτός ο σφιχτός αναγκαλισμός με την Ευρώπη. Έχουμε ανοιχτή αγορά, αλλά θα πρέπει να έχουμε και φύ μέτρα για να αποφύγουμε να δούμε οι αρχές αυτές της ανοιχτής Ευρώπης να χρησιμοποιούν τις βάρος μας. Έχω κάνει έξι τροπολογίες στη γνωμοδότηση του Τζέφρι Βαν και βεβαίως με χαρά προσβλέπω στην αυριανή συνάντηση και συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κλέρ Μόντι που είναι σκιώδης συζητήτρια εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Τζέφρι για την ε, γνωμοδότησή του αυτή που βέβαια συνεργαστήκαμε πάνω σε αυτήν με ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά σφιχτό. Οι σοσιαλιστές στηρίζουν λοιπόν τις προτάσεις που έγιναν. Αναγνωρίζουμε ότι προφανώς πολλά θετικά έχουμε από ξένες άμεσες επενδύσεις. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτές. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος των επενδύσεων. Να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει και ευθύνη για προστασία των βασικών υποδομών αλλά και των συμφερόντων μας κάθε φορά που εξετάζουμε τέτοιες επενδύσεις. δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει προστατευτισμό σε κάτι τέτοιο, όχι, αλλά πρέπει να παίρνουμε τις ευθύνες μας στα σοβαρά όταν πρόκειται για τέτοιες επενδύσεις. Η πρόταση τρέχουσα για παράδειγμα δεν κάνει καθόλου μνήα στην αμυντική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εξού και οι τροπολογίες μου αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτήν την απέτησή μας, να υπάρχει σαφώς μνήα της βιομηχανίας αυτής και του κλάδου αυτού. Η οποιαδήποτε πρόταση για αυτές τις επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικό έλεγχό τους. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εξετάζουμε τις ε, εξωτερικές άμεσες επενδύσεις. Να δούμε να λάβουμε υπόψη μας και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, κεφαλαίου. Τέλος. Ακόμα και αν έρχεται μια επιχείρηση από άλλα μέρη του κόσμου, και πάλι θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιες τρίτες χώρες ε, μπορεί να λειτουργήσουν με τρόπο που εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για ιδιωτικέ επιχειρήσεις. Οπότε πρέπει να δούμε τελικά από πού προέρχονται οι ξένες αυτές επενδύσεις. Πάντως, ευχαριστώ για την πρόταση και προσβλέπω στην αυριανή συνάντηση που θα έχουμε σκιώδεις συζητητές αύριο το απόγευμα για να καθίσουμε και να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες και έγκαιρα να τις έχουμε υποβάλει ώστε να μεταφραστούν κτλ. Ευχαριστούμε κυρία Άννα Ευχαριστώ. Χαίρομαι που φαίνεται ότι ξυπνήσαμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία και την χρήση στην άμυνα. Ευχαριστώ για αυτό που ακούσαμε πριν. Δηλαδή, να ζητάμε σε θελοντική βάση να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών δεν φτάνει για μένα. Χρειαζόμαστε επίσης μια καλύτερη χαρτογράφηση το από πού προέρχονται αυτές οι άμεσες ξένες επενδύσεις και να δούμε τις υποδομές και ποιος τελικά τις ελέγχει με τέτοιες υποδομές, με τέτοιες γνώμη επενδύσεις. Μην πως είναι ξένες δυνάμεις. Υπενθυμίζω στη χώρα μου, για παράδειγμα την Πορτογαλία, τη, στην εποχή εκείνη της νεοφιλελεύθερης εποχής που οδήγησε στη λιτότητα, οι υποδομές οι κοινοφελείς που αποδεσμεύτηκαν προκειμένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς, δηλαδή η διανομή και η παραγωγή της ενέργειας, διαχωρίστηκαν ακριβώς για να ισχύει ο ελεύθερος ανταγωνισμός όπως προβλέπουν οι κανόνες της εσωτερικής μας αγοράς. Ε, Υπήρξε επανασύνδεση όμως την εποχή της λιτότητας, τότε που είχαμε την Τρόικα, την Κομισιόν, δηλαδή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Εθνικό Νομισματικό Τομείο. Και ποιος έκανε αυτή την επανασύνδεση? Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Γιατί ήταν η κινέζικη εταιρεία η οποία επένδυσε για να ελέγξει την ε, παραγωγή ενέργειας στην Πορτογαλία και η κρατική λοιπόν κινέζικη τελικά εταιρεία είναι αυτή η οποία ελέγχει την παραγωγή ενέργειας στην Πορτογαλία. Παραγωγή ενέργειας έτσι που προφανώς και πρέπει να θεωρείται ένα κοινοφελές δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τα λιμάνια. Κοιτάξτε πόσα λιμάνια στην Ελλάδα και στη δικιά μου τη χώρα πουλήθηκαν αυτά τα χρόνια. Και έγινε συνειδητά αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέβλεψε. Ε, κλείνε τα μάτια μπροστά σε αυτά που πραγματικά συνέβαιναν. Όλα αυτά λοιπόν τα ήξερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν αυτή που τα επέβλεψε. Κρίσιμες υποδομές λοιπόν και βασικές επιχειρήσεις σε θέματα άμυνα, δεν ξέρω εγώ τι, τελικά αποξενώθηκαν από την Ευρώπη. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι άλλο. Δεδομένα, συλλογή δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες μέλη, πόσα από τα δημόσια τμήματα ελέγχονται τελικά από ξένες επιχειρήσεις, κινέζικες για παράδειγμα. Όλα τα δεδομένα δηλαδή, τα οποία θα έπρεπε να προστατεύονται, συλλέγονται και αποθηκεύονται που στην Κίνα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το Χαβέ είναι ένα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Δυστυχώς δεν ήμασταν έτοιμοι να συνειδητοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. σε ευχαριστώ. Ε, Πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει τον λόγο, κυρία Μπλάουερ. Καλησπέρα. Λίβια Πάουλερ, είμαι αναπληρωτής ε, ε, τμήματάρχης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω λίγο για το σχέδιο γνωμοδότησης αυτό που πήραμε κι εμείς. Ευχαριστούμε την Επιτροπή σας πρώτα απ' όλα για την γνωμοδότησή σας αυτή που μας στηρίζει και ευχαριστούμε που η γνωμοδότηση αυτή αναγνωρίζει την όλο και μεγαλύτερη ανησυχία μας όσον αφορά τις άμεσες ξένες ε, επενδύσεις στον τομέα των υποδομών και της άμυνας. Η συνεργασία επίσης αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία στην Ευρώπη και ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Και αναφέρεται και στη μελέτη μας όσον αφορά τη... το θέμα αυτό που δημοσιεύσαμε το 2017 σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα. Και σε μια πρόσφατη μελέτη της Egman που ονομάζεται «Κινέζικες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το σχέδιο γνωμοδότησης είδα ότι περιλαμβάνει μια ανησυχία. Λέει ότι η πρόταση ίσως ε, παραβαίνει πολύ στις αρμοδιότητες των χωρών μελών όσον αφορά την εθνική ασφάλεια και άμυνα. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι οι χώρες μέλη παραμένουν να έχουν το δικαίωμα εξαίρεσης που προβλέπεται από το συνδίκη όσον αφορά την ε, ε, από κοινού ενημέρωση, διαχείριση κλπ. δεδομένων. Η πρόταση αυτή λοιπόν δεν πλήττει αυτό το δικαίωμα. Υπάρχουν δύο τροπολογίες επίσης που έχουν ήδη εγκριθεί που μας ανησυχούν κάπως. Α, δεν έχουν εγκριθεί. Είναι δύο ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα. Ε, που προσέξαμε και μας προκαλούν κάποια ανησυχία. Η μία αφορά την, την κοινοποίηση περιπτώσεων που δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για την τροπολογία αριθμός 6, αν δεν απατώμε. Δεν θα είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση αυτή, αλλά σε θελοντική βάση. Κατά την άποψή μας αυτό αποδυναμώνει όμως την προστιθέμενη αξία που προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτή την πρόταση οι χώρες μέλη, εφόσον έχουν την επιλογή να το κάνουν ή όχι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ζητήσουν από την Κομισιόν ή άλλες χώρες ε, για γνωμοδότηση. Θα προτιμήσουν να το κρατήσουν για τους αυτούς τους. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι χάνεται πολύ προστιθεμένη αξία. Έπειτα, θα έπρεπε να περιορίσετε στην ασφάλεια η γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής και να μην αναφέρεται δημόσια τάξη. Επ' αυτού, για μας είναι δύσκολο μερικές φορές να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο, την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Η ασφάλεια προμήθειας φυσικού αερίου είναι υπό τη δημόσια τάξη και όχι υπό την ασφάλεια. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες μέλη να μπορούν να σχολιάζουν και όσον αφορά τη δημόσια τάξη. Έπειτα άκουσα κάποιον να λέει μήπως είναι πολύ λίγα όλα αυτά. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου 16 χώρες μέλη δεν κάνουν τον έλεγχο. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα δεν βλέπουν τις ίδιες ανησυχίες που βλέπετε κι εσείς. Υπάρχει ένα στοιχείο συνειδητοποίησης λοιπόν που θέλουμε να πετύχουμε με την πρόταση αυτή. Αν έπρεπε να επιβάλλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, αυτό σίγουρα θα υπερφόρτωνε την κατάσταση. Θέλουμε μια συνειδητοποίηση πρώτα. Και μετά, αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, και όχι ένα βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο, αλλά μακροπρόθεσμο, τότε θα εξετάσουμε παρετέρω Σε αυτό το στάδιο όμως πιστεύουμε ότι είναι μια ισορροπημένη πρόταση η οποία λαμβάνει υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στις χώρες μέλη υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να πάρω το λόγο μετά από μερικά από αυτά που είπατε. Ε, γιατί προέρχομαι από χώρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θεωρώ μάλλον θέμα ασφαλείας και όχι δημόσιας τάξης ε, την ε, προμήθεια φυσικού αερίου. Και πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου από την περιοχή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν μαζί μου. Ο κύριος Βαν Όρντεν, παρακαλώ. Για αυτό το τελευταίο σχόλιο σας, κυρία Πρόεδρε, ο καθένας, ε, ε, αν θέλει, μπορεί να ερμηνεύσει με την ευρία έννοια ε, το θέμα του δημοσίου συμφέροντος της δημόσιας τάξης και να εντάξει εκεί ό,τι θέλει. Εδώ φυσικά μιλούμε για θέματα ασφάλειας και η ασφάλεια βεβαίως εξορισμού είναι κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποιος έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τους συναδέλφους. Πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. Ακούω τα όσα λέτε και θα τα λάβω υπόψη μου και προσβλέπω και εγώ στην αυριανή μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, η γνωμοδότηση θα εγκριθεί το Μάρτιο, όπως είπαμε, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ στις 19 ε, ή 20 Μαρτίου όταν έχουν τη συνεδρίασή τους. Ωραία. Μην φύγετε σας παρακαλώ. Θα περάσουμε αμέσως μετά στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η 20 μαρτιου οταν εχουν τη συνεδριαση τους ωραια μη φυγετε σας παρακαλω θα περασουμε αμεσως μετα στο επομενο θεμα της Ευρώπης απέναντι στις ε, κυβερνοαπειλές. Περιμένουμε τα ξέχοντα μέλη του πάνελ. Ο κύριος Σολντάτοφ πρώτος έχει το λόγο. Colleagues, uh, Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο, όπως σας είπα, στη μέση διάταξη, είναι η προστασία της Ευρώπης εναντίον των κυβερνοαπειλών. Με μεγάλη χαρά, καλωσορίζω τους διακεκριμένους ομιλητές μας. Ένας εξ αυτών είναι Ρώσος, ρεπόρτερ, πολύ γνωστός, ο κύριος ε, Αντρέι Αλεξέιβιτς Σολτάτοβ, ο οποίος ηγείται μιας δουλειάς που γίνεται σε μια δικτυακή πύλη στα πλαίσια του Αγγεντούρα, ΔΟΤΡΟΥ, Είναι ένας δημοσιογράφος με εκτεταμένη πείρα, καλύπτοντας α, τις α, μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά αυτή στην α, Ρωσική Ομοσπονδία. Κάλυψε γεγονότα όπως τον Μπιουστράν και άλλες σημαντικές ιστορίες που συνέβησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία που ακόμα τις θυμόμαστε. Είναι γνωστός εμπειρογνώμονας για θέματα τρομοκρατίας, θέματα ασφάλειας. Θα θέλαμε να μας πει πολλά πράγματα Δυστυχώς πρέπει να σας περιορίσουμε όμως, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Πρέπει να περιοριστείτε στις ε, κυβερνοαπειλές. Και ένας ε, ανώτατος εκπρόσωπος του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ των ΗΠΑ, ο ο κύριος Μπρούνο Λετέ. Ο κύριος Λετέ θα παρουσιάσει πρώτος τις απόψεις του. Έχετε το λόγο, κύριε Λιτέ. Κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, ευχαριστώ και την Επιτροπή που με προσκάλεσε να την ενημερώσω. Μου ζήτησαν να ετοιμάσω την ε, συνεργασία, ε, κάτι για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για, την, ε, για θέματα άμυνας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τι συστάσεις έχω να κάνω εγώ για να προχωρήσουμε. Καταρχάς, τον κυβερνοχώρο, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι στόχος ε, των κυβερνοεγκληματικών, ε, μη κρατικών εταίρων για πολιτικούς λόγους και πολύ Προηγμένε ομάδε ομάδες και φορεί κτλ. Και, και αυτές οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της κοινωνίας της Ευρώπης ε, και του ΝΑΤΟ. Ε, πολιτική ασφάλεια, οικονομική, στρατιωτική κτλ. Παρότι οι επιθέσει στον κυβερνοχώρο είναι σοβαρέ απειλέ, οι καθημερινές ε, επιθέσει που γίνονται δεν τι παρατηρούμε, δεν τι ανοιχνεύουμε, δεν τι ξέρουμε ή εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζουμε ανεπαρκώς. Η κυβερνοασφάλεια και η άμυνα λοιπόν ε, επί μακρόν ήταν τμήμα των ε, υπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και μόνο πρόσφατα πέρασαν στο πολύ ψηλά στη μερίσια διάταξή τους. Η κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη ήταν το 2007 όταν έγιναν ε, στην Εστονία μεγάλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον της Εστονίας που ανάγκασαν και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτούν πιο σοβαρά το θέμα αυτό, αυτές τις απειλές. Ως αποτέλεσμα η Εστονία λοιπόν, ή τουλάχιστον εν μέρη, ε, το ΝΑΤΟ ε, δημοσίευσε το 2008 ε, την πρώτη του πολιτική για τις επιπλέσεις και πέντε χρόνια μετά το 2012 ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετώντα την πρώτη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Προχωράω λίγο στο 2014 η Ουκρανία μετά το, την επόμενη μεγάλη κρίση στην Ουκρανία λοιπόν η ρωσική ε, προσάρτηση της Κρυμαίας και τα λοιπά, τον Ντομπάς και τα λοιπά, ε, αυτά έγιναν μαζί με πολλές ε, κυβερνοεπιθέσεις παράλληλα. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και έκτοτε, από το 2014 και μετά δηλαδή, βλέπουμε ότι και οι δύο φορείς προσπαθούν να εναντικοποιήσουν τις πρωτοβουλίες τους στον κυβερνοχώρο. Δεν θα διατρέξω όλες τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι έχουν ήδη γίνει πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό για αυτή την ενημέρωση που σας κάνω είναι να πούμε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα έτσι κατεπήγοντος, ας πούμε, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησαν να συνειδητοποιούν ότι είναι συμπληρωματικέ δυνάμεις. Το πρώτο βήμα ήταν, ε, έγινε πριν από δύο χρόνια, το Φεβρουάριο του 2016, όταν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν μια τεχνική διευθέτηση για να βελτιώσουν τον επιμερισμό των πληροφοριών μεταξύ τους ε, και ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα Λίγου μήνε μετά, με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ του Ιουλίου του 2016 στη Βαρσοβία, ε, που δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για συνεργασία ε, ασφάλεια και άμυνα και και το, ε, συμπεριλαμβάνει και το κυβερνοχώρο εδώ. παρά την, τις πολιτικές αυτές συμφωνίες για συνεργασία, η πραγματική κυβερνοσυνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ είναι δύσκολη και οι θεσμικές επιλογές είναι συχνά πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν δύο, ε, λίγα βασικά ε, εμπόδια που θα ήθελα να υπογραμμίσω, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, υπάρχει μια έλλειψη ε, ε, ε επιμερισμού πληροφοριών. Ε, συχνά οι πληροφορίε αυτέ είναι διαβαθμισμένε, ε, και δεν υπάρχει κανάλι για να περάσουν αυτέ τι πληροφορίες προς το ΝΑΤΟ ή αντίστροφα μεταξύ των θεσμικών οργάνων Ευρωπαϊκή Ένωση. και ΝΑΤΟ. Και σε επίπεδο κρατών μελών συχνά τα κράτη είναι απρόθυμα να ε, μοιράσουν τις ε, απειλέ για την ασφάλεια. Επίσης, δεν υπάρχει ίδιο επίπεδο ετοιμότητα και αντοχή στον κυβερνοχώρο. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχουν όλοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό ας πούμε τιμότητας. Ε, γιατί συχνά στο, σε επίπεδο της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η εστίαση γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και παρά το ότι προσπαθούν να συντονίσουν τι εθνικές προσπάθειες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το αποτέλεσμα είναι περιορισμένο. Γιατί οι συστάσει του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τα κράτη-μέλη συχνά δεν είναι δεσμευτικέ. Και αυτό επηρεάζει φυσικά τα πράγματα. Ε, τρίτον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν κοινέ ε, κυβερνοασκήσει, ε, κατάρτιση και εκπαίδευση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Ε, στο, ιστορικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μόνο μία κοινή στρατιωτική άσκηση κάναν. Και αυτό είναι το 2003, που δεν είχε στοιχεία του κυβερνοχώρου. Ε, το Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ σχεδίασαν, αλλά δεν εφάρμοσαν περισσότερα γυμνάσια και ασκήσει το 2007, το 2010 και το 2014. Ακόμα και σήμερα, παρά την πολιτική όθηση που υπάρχει στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι αυτές οι ασκήσεις και τα γυμνάσια γίνονται χωριστά. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία για τους δύο εταίρους για να δημιουργήσουν μια κουλτούρα πραγματικής ε, εμπιστοσύνης και κατανόησης. Νομίζω λοιπόν ότι η προτεραιότητα για τον ΝΑΤΟ και την Ένωση είναι να βρουν συνένεση για το πώς θα κάνουν περισσότερα πράγματα μαζί μεγαλύτερη συνεργασία είναι πολύ σημαντική για να ε, αποτρέψουμε, να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε τις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και για να λογοδοτήσουμε βεβαίως όσοι τις διαπράττουν. Σε αυτή την επιτροπή θα ήθελα να κάνω λίγες συστάσεις λοιπόν για να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία. Καταρχάς, να σας πω ότι δεν εφαρμόζεται κατά ανάγκη από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά μπορεί να γίνει αν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείξουν το πραγματικό πολιτικό, έχουν το πραγματικό πολιτικό θάρρο και την επιθυμία να το κάνουν. Καταρχά να επιμεριστούν τι πληροφορίε του. Το, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΝΟ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κοινό κέντρο ανάλυση των κυβερνοαπειλών. Και οι δύο έχουν ε, αποδείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν σε κοινέ δομέ, παραδείγματο χάρη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστεία για την Αντιμετώπιση Κυβερνοαπειλών στο Ελσίνκι. Το να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κέντρο ανάλυση απειλών για τον κυβερνοχώρο μεταξύ των δύο θα ήταν ένα επόμενο βήμα ε, για τη θεσμική συνεργασία των δύο. Και αυτό το κέντρο θα διευκόλυνε την ε, επίσημη και άτυπη ε, τακτική, ε, έτσι, τον τακτικό επιμερισμό πληροφοριών ε, μέσα από ασφαλείς διάβλους επικοινωνίας και έτσι θα ξέρουμε πότε θα επιμερίζονται, θα τις επιμερίζονται αυτέ τι πληροφορίε κτλ. Θα μπορούσαν να έχουν επίσης μια κοινή ομάδα εργασία για να συγχρονίσουν τα συστήματα απόκρισης τη κρίση. Σήμερα ε, ο μηχανισμός απόκρισης δεν είναι συντονισμένος ανάμεσα στου δύο και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα για να αποκριθούν από κοινού σε κυβερνοεπιθέσει. Μια κοινή ομάδα αυτή ε, θα γεφύρωνε το χάσμα και τελικά θα δημιουργούσε ε, ένα εγχειρίδιο ε, για το πώς αντιμετωπίζαν τις κρίσεις ε, οι δύο. Επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε ασκήσεις κοινέ για την κυβερνοασφάλεια και άμυνα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. σήμερα δεν υπάρχουν τακτικά οργανωμένες ασκήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αλλά για να καταλάβουμε ως τον άλλον. αν το κάναμε, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, και να μπορούμε τελικά να μοιραζόμαστε πληροφορίες. Τέταρτον, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές ε, για τον κυβερνοχώρο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ε, για να συμπεριλάβουμε απειλές ε, που αφορούν εξωτερικούς, που προέρχονται από εξωτερικούς αντιπάλους. Αν δείτε τι κάνουμε σήμερα, είμαστε, ομφαλοσκοπούμε γύρω από τις, τις δυνατότητες των κρατών μελών ε, οι, οι αντίπαλοι μα ε, επιτίθενται με βάση τα δικά μα ευάλωτα σημεία. Παραδείγματο χάρη τα ανεργά μέτρα, όπω λέμε, τη Ρωσία, που έχουν σαν σκοπό να εκμεταλλευτούν τις ε, τα σημεία που είναι ευάλωτα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ε, προσαρμόζονται οι ρωσικές δυνατότητες ε, μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο συμβατικών, υβριδικών και πυρηνικών δυνατοτήτων. Ε, επομένως, θα πρέπει να έχουν μια προσέγγιση ανοιχτή προς τα έξω, να μελετούν αυτές τις στρατηγικές και, το, τις δυνατότητε των αντιπάλων και να προσαρμοζόμαστε. Θα πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί για να αποτρέπουμε καλύτερα και να ε, αντεπιτιθέμεθα στις κυβερναυτές επιθέσεις. Πέμπτον, πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με, τα, με τους συνεργάτες μας. Καταρχά, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΝΑΤΟ. Αλλά είναι και το πρώτο, θα μπορούσε να είναι και το πρώτο ρήγμα. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθίσουν όλου του εταίρου του πιο ανθεκτικού, ούτω ώστε να κερδίζουν όλε οι πλευρέ. Ε, οι χώρε εταίροι θα πρέπει να ενισχύσουν το τεχνικό κύβερνο δυναμικό του και τα δίκτυά του και τα επίπεδα τα επίπεδά τους και οι εταίροι μας αυτοί θα μπορούν σε θέση να επιμερίζονται αυτές τις πληροφορίες στην πραγματογνωμοσύνη. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ε, συλλογική κυβερνοασφάλεια και άμυνα. Ε, ένα κοινό Trust Fund Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ για το κυβερνοχώρο θα μπορούσε να δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσουμε ε, και να εκμεταλλευτούμε τι δεξιότητε τις δεξιότητες που υπάρχουν και να επιτρέψουμε στους εταίρους να παραστούν, ας πούμε, σε, να, να παρίστανται σε σεμινάρια, εκπαίδευση κτλ. Ε, τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να πιέσουν και μια διεθνή συνεργασία που θα ε, ρυθμίζει την κρατική συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο. Ε, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι τα πρώτα θύματα όλο και περισσότερο των κυβερνοαπειλών. Κοιτάξτε, ας πούμε, τις επιπτώσεις. Ας πούμε, ε, στα οικονομικά μας συστήματα και στο σύστημα υγείας. Ε, αν δεν υπάρχουν ε, διεθνείς ε, συμβάσεις κτλ. δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς κυβερνοαπειλές της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξουν ηγετικό ρόλο για να προωθήσουν προτάσεις που θα προστατεύουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να ρυθμίζουν την συμπεριφορά των κρατών στον κυβερνοχώρο. Αυτό μπορούν να το κάνουν υποστηρίζοντας τις ισχύουσες πρωτοβουλίες σε επίπεδο G7 ή ΟΗΕ, αλλά να δούνε και τις ιδέες που υπάρχουν από άλλους τομείς, παραδείγματος χάρη τον ιδιωτικό το, τομέα, ας πούμε, ε, για να ενισχύσουν την ε, λογοδοσία και τη διαφάνεια. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το βασικό μου μήνυμα είναι η ανάγκη να προσαρμοστούν ο ένας τον άλλον, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες πιέσεις, ε, πέρα από τις παλιές προβληματικές ε, σχέσεις ε, που υπάρχουν εδώ και χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίσουν νέες κυβερνοαπειλές. Παρόλα αυτά σήμερα ακόμα είναι ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο περιβάλλον για την ασφάλεια. Η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να δείξει ότι είναι αξιόπιστη στον κυβερνοχώρο ως μια ισχυρή δύναμη στα μάτια των μελών, εταίρων και αντιπάλων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αντρέι Σολτάτοφ τώρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε και για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Όλοι, όταν σκεφτόμαστε απειλές στον κυβερνοχώρο, σκεφτόμαστε τη Ρωσία για προφανείς λόγους και υπάρχουν προφανείς λόγοι γι' αυτό. Και ένα πράγμα που θα ήθελα εδώ να σας πω είναι ότι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, γιατί ε, προχωρούν με αυτόν τον τρόπο στον κυβερνοχώρο οι Ρώσοι που είναι μοναδικός. Πράγματι, μιλάμε για την ασφάλεια. Είναι εντελώ διαφορετικό αυτό που υπάρχει στη Δύση με αυτό που υπάρχει στην Κίνα, για παράδειγμα. Και Μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Οι Ρώσοι που κάνουν τις απειλές αυτές στον κυβέρνο χώρο είναι επιτυχείς εκτός της χώρας, ενώ μέσα στην ίδια τη Ρωσία δεν ε, τα καταφέρνουν. Έχουμε ακόμα μια επιλογή που μπορεί ο κόσμος online να εκφράζεται και έχουμε και δυνατότητα να βγαίνει ο κόσμος στο δρόμο, ή να διαδίδει πληροφορίες παρά τις όποιες κυρώσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο. Εκτός της χώρας όμως οι άνθρωποι αυτοί τα καταφέρουν καλύτερα και αυτό θα έπρεπε να έχει κάποια εξήγηση. Το άλλο είναι ότι όταν μιλάμε για τον κυβερνοχώρο μιλάμε συνήθως για ένα συγκεκριμένο παράγοντα, σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Με την περίπτωση της Ρωσίας είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Μιλάμε για κρατικούς παράγοντες, επίσης για επίσημους παράγοντες, αλλά και για μη κρατικούς. Είναι πολύ περίπλοκη η σχέση μεταξύ των στρατιωτικών στη Ρωσία και την ασφάλεια, των Ρώσων hackers, ε, ε, των επιχειρήσεων πληροφορικής στη Ρωσία. Κάτι άλλο είναι. Έχω την εντύπωση ότι όταν η Δύση προσπαθεί να μιλήσει με επίσημους φορείς της Ρωσίας, Τελικά είναι σαν να μιλάνε με λάθος ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να φαίνεται ότι είναι επίσημοι με όλα τα διαπιστευτήρια κτλ. Αλλά τελικά δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Και έπειτα η λεγόμενη chain of command. Λέμε ότι μιλάμε με μια χώρα η οποία είναι γνωστή ε, ως μεγάλη, αποκεντρωμένη, με μία με πολύ, που δεν είναι αποκεντρωμένη, που είναι, έχει μια πολύ συγκεντρωτική δίκηση, όμως τελικά δεν έχουμε ιδέα για το πώς γίνονται κυρώσει, αν γίνονται κυρώσει, από πού κατευθύνονται αυτές. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα και θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί η ρωσική προσέγγιση όσον αφορά το κυβερνοχώρο έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί ένα ιστορικό. Πώς θα έπρεπε να το δούμε. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε για ένα στρατηγικό σχέδιο της δεκαετίας του 80 ή του 90. Εδώ πρόκειται για τακτικής φύσεως αποφάσεις μετά από κρίσεις. Η πρώτη κρίση ήταν στο Κρεμλίνο εξαιτία του πολέμου στη Τσετσενία. Όχι μόνο γιατί επρόκειτο για μια μετοχυσία, στρατιωτικού τύπου, αλλά για το 99, το 2000 χρειαζόταν μια εξήγηση το Κρεμλίνο γιατί να πάει στο δεύτερο πόλεμο και έπρεπε να το πουλήσει αυτό στον πληθυσμό. Και άρα έπρεπε να εξηγήσει και γιατί χάσανε τον πρώτο πόλεμο. Η εξήγηση ήταν ότι χάσαμε τον πρώτο πόλεμο εξαιτία τη δημοσιογραφία, εξαιτία τη πληροφόρηση τότε ήταν που άρχισαν να αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες και την ενημέρωση σαν ένα εχθρό. Από τα διάφορα έγγραφα που έχουμε είναι ολοφάνερο ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας θεώρησαν σαν όπλο την ε, πληροφόρηση και τους δημοσιογράφους τους αντιμετώπιζαν σαν ενδυνάμει επικίνδυνους που θα έπρεπε να δρανοποιηθούν. Όμως χάσανε. Ήταν σαν να μιλάμε για ε, λογοκρισία. Και βέβαια και υπάρχει λογοκρισία, αλλά όχι μόνο. Ήταν και θέμα κυβερνοχώρου. Γιατί όταν ε, έχετε αδρανοποιήσει τους δημοσιογράφους σας, υπάρχει πάντα το διαδίκτυο. Οπότε οι αποσχιστές ε, Τσετσένοι είχαν ε, ιστοσελίδες σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ρωσία, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν κατάφερε να πείσει τις δυτικές χώρες να κλείσουν τις ιστοσελίδες αυτές. Υπήρξαν ε, φοιτητέ στην Σιβηρία, στο Τόμσκ, που από μόνοι τους είχαν ιστοσελίδα. Και οι τακτικές ε, αυτές του outsourcing έτσι γεννήθηκαν. Κάποιοι απλώς έπρεπε να ενθαρρυνθούν ή να κατευθυνθούν κατά κάποιων στόχων, ακόμα και αν δεν είναι κρατικοί παράγοντες. Τέτοιες τακτικές λοιπόν έχουν αναπτυχθεί πολλοί. Φοιτητέ, κινήματα νέων, hackers, εγκληματίες και η τάση αυτή μεγαλώνει. Η ιδέα πάντως ότι ακόμα και αν έχετε κάποιους Ρώσους hackers αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάτε για την κυβέρνηση και ότι πάντα μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι δικιά σας ευθύνη και να πείτε κάποιος άλλος το έκανε, δεν το έκανε η κυβέρνηση, παραμένει ως ε, δόγμα. Και ακριβώς περί αυτού πρόκειται τώρα. Και το πρόβλημα είναι ότι ασφαλώς και δημιουργείται έτσι μία αίσθηση νομίζω ότι είσαι υπό επίθεση, αλλά δεν υπάρχει στρατηγική για να απαντήσεις. Και η ότι μπορείς με τέτοια όπλα εξίσου να αντιμετωπίσεις τέτοιες επιθέσεις δεν ισχύει, γιατί δεν έχει τέτοια μέσα όπως έχουν οι Ρώσοι. Τα CBS, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι Αμερικανοί το είχαν προτείνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Θέλανε να μιμηθούν αυτό που υπήρχε τη δεκαετία του 70 και του 80 μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, ότι άπαξ και υπήρχε μια κρίση, σήκωνε το τηλέφωνο ο πρόεδρος, μιλούσε με τον ομολογό του, του έλεγε να έχουμε εδώ πέρα κάτι με τους πυράβλους, για επιβεβαίωση αυτό, τι θα κάνουμε μετά. Αυτή η κόκκινη γραμμή λοιπόν υπήρχε ήταν κάτι γνωστό και προσπάθησαν να την επανεργοποιήσουν το 2016. Αλλά δεν πέτυχε γιατί ο αρμόδιος του Ομπάμα έκανε ε, το τηλεφώνημα αυτό, αλλά από πλευρά τη Ουάσιγκτον υπήρξε πλήρη σιωπή. Και γιατί? Από πλευρά τη Ρωσία, συγγνώμη, υπήρξε μια πλήρη σιωπή. Θα πρέπει να υπάρχει νέα προσέγγιση τώρα. Όταν ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η δυσπιστία, υπάρχει και μεγάλη τάση να προσπαθήσει κανείς να στρατικοποιήσει το θέμα. Ανάμεσα των Ρώσων αξιωματούχων και των Δυτικών αξιωματούχων πάντα υπήρχε διαφωνία για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα του κυβερνοχώρου. Για δεκαετίες οι Ρώσοι θέλαν να μιλήσουν για την ασφάλεια της πληροφορίας, ενώ από την άλλη μεριά θέλω να μιλήσω για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το πρώτο έχει να κάνει με το, με το περιεχόμενο, ενώ η δυτική προσέγγιση είχε να κάνει με την πληροφορική, τους υπολογιστές. Και έτσι τα τελευταία χρόνια και στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο μου λένε κατά πάσα πιθανότητα δίκιο είχαν οι Ρώσοι. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για την ασφάλεια του περιεχομένου. Αυτό θα ήταν επικίνδυνο. Πρώτα απ' όλα ως δημοσιογράφος, εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος με τη γνώμη ότι η πληροφορία είναι ένα όπλο. Είναι επικίνδυνο αυτό. Ενώ αν περάσουμε σε αυτή την ιδέα, τότε με τον άλλο με τον άλλο τρόπο θα καταλήξουμε σε λογοκρισία. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η ιδέα της στρατιωτικοποίησης του θέματος είναι κάτι πολύ δυτικό. Στη Ρωσία πάντα για 20 χρόνια και ήταν θέμα των υπηρεσιών ασφάλειας στη Ρωσία και όχι των στρατιωτικών. Όταν χωρίστηκε η Καγκεμπέ, το ένα κομμάτι της ΚΑΚΕΜΠΕ πήρε αυτό το ζήτημα και όχι οι στρατιωτικοί, οι οποίοι αποκλείστηκαν από αυτό για πολύ καιρό. Η Δύση όμως ήθελε τη ρωσική προσέγγιση να την αντιμετωπίσει σαν κάτι συγκρίσιμο με τη δυτική προσέγγιση. Και επειδή στη Δύση υπήρχε σχέση και με το στρατιωτικό σκέλος, δεν μπόρεσε αυτό να λειτουργήσει. Πρόκειται για διαφορετικούς φορείς, για διαφορετικές στρατηγικές και για διαφορετικές ιδέες. Όταν όμως μιλάμε για την στρατιωτικοποίηση, το πρόβλημά μου είναι ότι μπορεί να καταλήξετε σε λογοκρισία. Γιατί αυτό κάνετε όταν έχετε πόλεμο, έτσι δεν είναι. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι το πραγματικό θέμα εδώ δεν είναι να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όρους πολέμου, αλλά να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τους ανθρώπους που προχωρούν σε πράξεις που θεωρούνται παράνομες σύμφωνα με την νομοθεσία διάφορων χωρών. Και αυτό το είδαμε όταν βγήκε η δικαστική απόφαση για το Μίλλερ. Και τελικά θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οργανώνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί η απόφαση για το Μίλλερσον, για παράδειγμα, μας έδωσε μια εικόνα για το πώς λειτουργούν αυτά τα ζητήματα. Έχετε όλους αυτούς τους άτυπους φορείς. Παρ' όλα αυτά έχετε την εικόνα Αυτό μπορεί να αποφέρει καρπούς. Τέλος. Το να θεωρούμε την πληροφόρηση σαν ένα όπλο. Είναι ο ρωσικός τρόπος να αντιμετωπίζει τον κυβέρνο χώρο. Γιατί στο Κρεμλίνο πολλοί προέρχονται από την ΚΑΚΕΜΠΕ και έχουν καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουν τον κόσμο ως μια απειλή. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Δεν πρόκειται μόνο για απειλή. Το διαδίκτυο προσφέρει πάρα πολλές ε, ευκαιρίες σε όλους. Όλοι περνάνε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι πολύ υποσχόμενο. Δεν πρόκειται μόνο για μια απειλή και για κάτι επικίνδυνο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει λοιπόν τώρα η συζήτηση. η κυρία Μόντι, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Έχω δύο ε, σχόλια και για τους δυο σας. Το πρώτο αυτό που αναφέρατε για την ε, διακήρυξη της Βαρσοβίας και τη συμφωνία του 2016 για το τι χρειάζεται να γίνει, που το αναγνωρίσαμε εκεί, αλλά δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα σχέδια και να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση ε, ώστε να αποδώσει. Υπάρχει μια τάση εδώ που έχουμε εμείς, ε, έτσι, σπέρδευρα δέος. γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει για τον τελικό μας προορισμό. Συμφωνείτε με αυτό. Αυτό τώρα τι είναι, ραστόνι, βραδιπορία, τι πρέπει να κάνουμε, ποια θα ήταν τα καλά βήματα για να έχουμε αποτελέσματα. Ε, με αυτό τον τρόπο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ εννοώ να έχουμε ένα ασφαλή χώρο για αυτή τη συνεργασία. Κύριε Σολντάτοφ, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και θέσατε ένα θεμελιώδες ερώτημα, που είναι το ζήτημα του περιεχομένου. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να ανοίξει ε, ε, ο χώρας να τον ανοίξει για τη λογοκρισία είναι το αντίθετο αυτό που θέλουμε. Ε, πραγματικά εκεί είναι το πρόβλημα, το περιεχόμενο και το θέμα της παραπληροφόρησης και όχι της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Πριν ε, αυτό το πρόβλημα. Γιατί βλέπουμε να λιώνεται όχι μόνο η πληροφόρηση, αλλά η ίδια η γλώσσα. Το έχουμε δει στη χώρα μας αυτό όλοι, στις διάφορες χώρες μας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το περιεχόμενο και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ε, ξεφύγουμε από εκεί και να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα φαίνεται ότι δεν είμαστε στο ύψος περιστάσεως για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Ε, θα θέλαμε να το διερευνήσουμε λίγο περισσότερο. Τι θα κάνουμε το περιεχόμενο. Χωρίς να μπαίνουμε στη λογοκρισία, αλλά οπωσδήποτε αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Mr. Tune Ο κύριος Τούνε Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ εύστοχα και, και χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Μούντι είναι υψή σημασία στο θέμα του περιεχομένου. Και η ρωσική πλευρά και γενικότερα τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν στρατηγική στην προοπτική τους. Εμείς απλώς αντιδρούμε. Έχουμε διαφορά στην αντίληψη και στον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας μας. Ταυτόχρονα όμως ανησυχώ λίγο, διότι το κοινοβούλιο μας ενέκρινε την πρώτη έκθεσή του για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πριν από 5-6 χρόνια τουλάχιστον. Και τα θέματα, αυτά τα ίδια θέματα ε, ήταν ε, στην έκθεση αυτή. Η ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η συνειδητοποίηση των κρατών μελών, τιμότητα των κρατών μελών, ζητήματα που έχουν να κάνουν με συνεργασία ιδιωτικού με δημόσιο τομέα, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ε, hackers που δεν ε, εκπροσωπούν κράτη. Πρόσφατα τα κράτη-μέλη άρχισαν και εκείνα να χρησιμοποιούν τους hacker ε, θετικούς για, να αποκρούσουν αυτές τις επιθέσεις, για να αντιπιθύνται. Έχουμε τους καλούς hacker τώρα εμείς. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Υπάρχει ένα κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ για την ανάλυση των απειλών στον κυβερνοχώρο. Ε, αυτό προτείνεται ως ιδέα. Αυτό που έχουμε στο Ταλίν θα μπορούσε να αποτελέσει βάση. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα παράλληλο κέντρο, διευρυμένο κέντρο και για να το σκοπούς. Σε τελική ανάλυση, το θέμα είναι να έχουμε συνειδητοποίηση, επαγρύπνηση και έπεται η πολιτική βούληση για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Και όχι απλώ ωραία λόγια και διακήρυξει, αλλά και να μπούμε στην πρακτική συνεργασία. Η ανάλυση σας είναι πάρα πολύ ρεαλιστική κατά την άποψή μου. Χρειάζεται να δοθεί συνέχεια αλλά το αιώνιο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Γκόμες. Thank you. Um, I, I took note of the very... Κατέγραψα τις ε, σημαντικές ε, προτάσεις του κυρίου ΔΕΤΕ για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τα ευάλωτα σημεία που έχουν στον κυβερνοχώρο. και αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοαπειλές. Η συνεργασία όμως των δύο πάντα εμποδιζόταν από πολλούς παράγοντες, κυρίως θέμα της ε, Τουρκίας-Κύπρου, τέτοιου τύπου προβλήματα. με διαφορετικά αφηγήματα για το που πάμε. Στο σημερινό κόσμο το... ο κυβερνοχώρος περιπλέκει τα πράγματα και τις σχέσεις. Το ίδιο θα μπορούσα να πω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο βασικός ε, εταίρος του ΝΑΤΟ, όμως με το νέο πρόεδρο, ε, μην ξεχνάω ότι γίνεται μια έρευνα εναντίον του πρόεδρου για τις σχέσεις που έχει αυτή η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρόεδρος, οι στενοί του συνεργάτε με τη Ρωσία. Αυτό ισχύει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν βοηθάει βεβαίως. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι λόγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην κάνει τίποτα. Αντίθετα, θα πρέπει να προχωρήσει με ή χωρί το ΝΑΤΟ. Και τώρα ας περάσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σολντάτοφ. Συμφωνώ μαζί σας ότι η πληροφορία δεν είναι όπλο, αλλά χρησιμοποιείται ως τέτοιο. Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ε, αυτό το γεγονός και να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Όχι με τη χρήση των ίδιων πυρομαχικών, αλλά δείχνοντας ότι δεν είμαστε αφελείς και ηλίθιοι και δεν επιτρέπουμε να μας πλήξουν αυτά τα όπλα. Το όπλο αυτό της ε, πληροφορίας, των πληροφοριών ή της ενημέρωσης. Γιατί χρειαζόμαστε την, ε, το RT και το Sputnik ε, εφόσον έχουμε το Euronews. Το Euronews ε, το πληρώνουμε 30 εκατομμύρια ε, το χρόνο, αλλά δεν ελέγχει το περιεχόμενο. Εγώ δεν θέλω να ελέγξω το περιεχόμενο, αλλά την, να είναι αποτελεσματικό. Να μην είναι, ας πούμε, εργαλείο ε, προπαγάνδα στο Euronews για τον Πούτιν, ας πούμε. Ή για το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν, ας πούμε. Ή ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε πραγματικά τα γεγονότα. Ε, state or non-state. Για το τι κάνει ας πούμε το Russia Today ε, ή ρωσικη ρωσικοί κρατική και μία ας πούμε και να ξέρουμε τι είναι fake news και τι όχι. Κύριε Σολτατόφ, νομίζω το πιο σημαντικό εργαλείο σήμερα που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για την άμυνά μα και την ασφάλεια για να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνοαπειλέ, είναι να δείξουμε τη διαφθορά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσω του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, μέσω ερευνών, από ρεπόρτερ όπως ο Κρουσόσορ που ε, δημοσίευσαν τα έγγραφα του Παναμά και τα Paradise Papers. Τι νόημα έχει Ας πούμε ο κύριος Μπουζεμπάουερ υποστήριζε το καθεστώς ε, Γιανουκόβιτς. Ήταν ο πιο θερμός ε, υποστηρικτής του από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δεν ήταν ο μόνος, φυσικά υπάρχουν και άλλοι υποστηρικτές. Το θέμα λοιπόν ε, καταπολέμησης της διαφθοράς και το, το να δείξουμε ποιοι είναι οι διεφθαρμένοι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την άμυνα. Ε, τίποτα δεν είναι πιο αποτελεσματικό από τους ε, δημοσιογράφους, στον κυβερνοχώρο μάλιστα, που με τα εργαλεία αυτά όπως τα Panama Papers και τα Paradise Papers ας πούμε, εξέθεσαν αυτή τη διαφθορά, παρουσίασαν αυτή τη διαφθορά. Πολλές από τις πληροφορίες στα Panama Papers ε, ε, υπέδειξαν ότι από πίσω είναι ο Πούτιν και η δική του και που ξέπλαιναν χρήματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο, και αλλού ας πούμε, αλλά μέσω διαφόρων ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Κύπρος, η Μάλτα, οι μικρές αυτές χώρες, αλλά είναι και η Ολλανδία, η Αυστρία, το Λονδίνο. Πολύ. Αυτά τα ξέρει η ρωσική κοινή γνώμη. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να αντιμετωπιστεί αυτή η προπαγάνδα, για να καταλάβουν οι Ρώσοι τι παίζεται εδώ, ε, οι δικοί τους ας πούμε, οι διεφθαρμένοι ας πούμε, elite, τι κάνουν. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Οι ερωτήσεις. Μία προς τον κύριο Σολντάτοφ. Ποια είναι η φύση των, του τρόλινγκ στο κυβερνοχώρο στη Ρωσία. Πώς γίνεται το τρόλινγκ εγώ έπεσα θύμα πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι το κάνουν πολύ καλά. Και το κάνουν πολύ καλά σε, σε ορισμένε χώρες να παρεμποδίζουν μηνύματα, να μπλοκάρουν μηνύματα, ας πούμε. Που αν διαδιδόταν δεν θα ήταν επωφελή για τη Ρωσία. This area is quite well organized and, quite effective. It's not only students. Νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικά οργανωμένα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το, το hacking δεν το κάνουν μόνο οι, οι φοιτητέ. Υπάρχει ένα στρατό από ανθρώπους που μπλοκάρουν τα θετικά μηνύματα της δύση από το να κυκλοφορήσουν εντός της Ρωσίας. Μπρούνο Λετέ. Μετά τη συνοκορφή της Βαρσοβίας, το θέμα της κυβερνοασφάλειας μπήκε ψηλά στην ατζέντα. Ένα είδος πολέμου θεωρήθηκε ότι είναι. Γίνεται εκεί στο ίντερνετ. Και διάφοροι σύμμαχοι μας αποφασίσαμε ε, να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε πιθανές επιθέσεις που θα μπορούν και στρατιωτικού χαρακτήρα. Τι μπορούμε να κάνουμε η μεν και η δε μπορεί το ΝΑΤΟ να συμπληρώσει τη δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστροφα. Πώς μπορούμε να διαιρέσουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Μια και το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει τη συλλογική μας άμυνα. Και η ΚΠΑ εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, αλλά με διαφορετική εστίαση από το ΝΑΤΟ που εξασφαλίζει τη συλλογική μας άμυνα. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία σε στρατιωτικό και μη σκέλος. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. να απαντήσετε με την ίδια σειρά. Ο κύριος Λεβέ πρώτα και μετά ο κύριος Σολτάδο. Παρακαλώ. Ο κύριος Λετέ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ερωτήσεις σας, για τα σχόλιά σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Στην κυρία Μούντι πρώτα απ' όλα. Ο κυβερνοχώρος είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει όταν σκέφτομαι τη συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή η συνεργασία πάει πολύ καλά. Σίγουρα γνωρίζετε ότι η κοινή δήλωση ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τέσσερις τομείς συνεργασίας είναι πώς θα η υπόψη ο κυβερνοχώρος, δηλαδή και οι σε αποστολές και επιχειρήσεις, η εκπαίδευση, κατάρτιση, οι ασκήσεις και τα πρότυπα. Η συνεργασία αυτή, λοιπόν, είναι από τα πράγματα που λειτουργούν καλύτερα όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Παραμένουν όμως προκλήσεις. Όπως είπα, Το θέμα είναι ότι παρά το γεγονό ότι έχουν εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να συντονίζουν τις προσπάθειες των χωρών μελών σε εθνικό επίπεδο, ο κυβερνοχώρος, η ικανότητα στον κυβερνοχώρο ή της πληροφόρησης παραμένει λεπτό θέμα για πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για πολλούς και διάφορους λόγους. Η της πληροφορηση παραμενει λεπτο θεμα για πολλες ευρωπαικες πρωτευουσες για πολλους και διαφορου λογους η εντολη ετσι κι δεν είναι δεσμευτική. Οπότε συχνά οι χώρες μέλη δεν θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν με άλλες πρωτεύουσες ή με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στις Βρυξέλλες. Πώς μπορούμε να τις κάνουμε να νιώσουν ότι έχουν κίνητρο για να το κάνουν όμως αυτό. Θα μπορούσαμε δείχνοντας τα θετικά, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε για να το πούμε αυτό. Οπότε τι θα πρέπει να κάνουμε τι, ποιος είναι ο στόχος μας. Δηλαδή, λέμε σε πέντε χρόνια ή του χρόνου, πού θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Για να δείξουμε ότι υπάρχουν αυτά τα κίνητρα. Μπορούμε να πετύχουμε καλύτερο έλεγχο. Ε, μπορούμε να έχουμε εκθέσεις πρόδου. Όχι να δείχνουμε με το δάχτυλο αυτόν που δεν τα έκανε καλά. Naming and shaming. Όχι, δεν λέμε αυτό. Η ρεαλιστική μέθοδος είναι αυτό να γίνεται σε θελοντική βάση. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στις χώρες μέλη αυτή τη συνεργασία. Αλλά να υπενθυμίζουμε πόσο πολύ επήγε αυτή η συνεργασία. Τώρα για την ερώτηση του κύριου Κέλαμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κέντρο αριστείας στο Ταλίν βοηθάει. Είναι όμως ένα ανεξάρτητο κέντρο αριστείας, το οποίο θεωρητικά δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει επίσημα θεσμοθέτηση αυτής της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ με τις διάφορες πρωτεύουσες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ ώστε να φανεί αυτή η σχέση και έτσι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τις διάφορες πρωτεύουσες, οι οποίες να προσφέρουν πληροφορίες και να διευκολύνουν τον επιμερισμό τους. Αυτό θα έπρεπε να είναι το κεντρικό σημείο. Το κέντρο αυτό στο Ταλίν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πράγματι. Αλλά αυτό που κάνουν είναι πραγματογνωμοσύνη, κατάρτιση και κατά την ταπεινή μου γνώμη θα ήταν προτιμότερο να είχαμε ένα κέντρο το οποίο θα έχει σαν αποκλειστική αρμοδιότητα τον επιμορισμό των πληροφοριών. Για να μην ξεχάσω τώρα τις ερωτήσεις σας, να δω... Α, κυρία Γκόμες, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας για την ερώτησή σας. Ναι, συμφωνώ με τις ανησυχίες σας για τον προβληματισμό όσον αφορά την Τουρκία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε με έρευνε, ναι, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά να ξέρετε ότι το αμερικανικό σύστημα δεν περιορίζεται στο λευκό οίκο. Ε, υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν στην διάρθρωση και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ δεν έχουν αλλάξει μετά την έλευση του τελευταίου Πρόεδρου. Προς το παρόν τουλάχιστον αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα θα έπρεπε να προχωρήσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι η απάντηση. Θα έπρεπε και ελπίζω στο πλαίσιο που προσφέρει η ΠΕΣΚΟ. Ίσως εκεί η διάσταση του κυβερνοχώρου να μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο. Και επίση από τα επενδυτικά ταμεία, μήπως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και προπολογισμό για την ικανότητα όσον αφορά το κυβερνοχώρο στις διάφορες χώρες, που θα πρέπει να ενισχυθεί. Η ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει προφανώς και ισχυρό ΝΑΤΟ. Είναι πράγματα συμβατά μεταξύ τους. Όσον αφορά τις δικές σας ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κυρία Φωτίγκα, είναι περίπλογο και νομίζω ότι κάθε οργανισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ διαθέτουν μοναδική πραγματοσύνη. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα που μπορεί να κάνει καλύτερα το ΝΑΤΟ. Πάντως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, καλύτερη συνεργασία. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όταν μιλάμε για ρυθμίσεις, για εμπόριο, για μη στρατιωτική χρήση. Το ΝΑΤΟ από την άλλη μεριά πρέπει να επικεντρωθεί στην ασφάλεια και την άμυνα, που είναι πράγματα που τα γνωρίζει καλύτερα. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τάση στο ΝΑΤΟ τώρα, στη Συμμαχία φαίνεται, ότι είναι πιο ανοιχτό για να μιλήσει για η ικανότητα στον κυβερνοχώρο πιο επιθετική, κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο πριν από ένα χρόνο. Αλλά η συμμαχία γίνεται πιο ανοιχτή και σε αυτή την επιλογή, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, και πάλι, για την διάκριση που δεν είναι σαφής, ναι, αλλά όσο προχωράει η συνεργασία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τις αρμοδιότητες καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Σολτάτοφ. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Να αρχίσω από την τελευταία, κυρία Φωτίγκα, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικό παράδειγμα. Γιατί είναι τόσο μοναδική η ρωσική περίπτωση. Υπάρχουν κάποιοι άτυποι ενεχόμενοι, όχι μόνο φοιτητέ, ε, και κάποιοι άλλοι που δεν συνδέονται ούτε με τη γραφειοκρατία, ούτε με τη διοίκηση, ούτε με το Κρεμλίνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι οργανωμένοι, ότι δεν είναι καλά οργανωμένοι. Uh, Ο μόνος ε, ε, ε, λόγος, μάλιστα από το 2005-2006 έχουν αρχίσει τα ρωσικά τρόλ. Ε, χρόνια ολόκληρα, γιατί η ρωσική γραφειοκρατία ε, είναι γνωστή για τη βραδύτητά της και οι μυστικές υπηρεσίες και όταν γνώρισε κρίση το Κρεμλίνο και θέλαμε να τη λύσουμε πολύ γρήγορα με το διαδίκτυο, εκείνοι απευθύνθηκαν ακριβώς σε άτυπους φορείς, ε, διότι θεώρησαν ότι είναι πιο αποτελεσματικοί. Πράγμα που αποδείχτηκε όντως. Για ποιο λόγο, διότι εκεί δεν χρειάζονται κυρώσεις. Είναι σε άμεση σύνδεση με το Κρεμλίνο, ξέρουν να ανοίξουν τις σωστές πόρτες Και πρόσφατα ε, ο Μιούλερ δημοσίευσε ε, ε, μια εργασία για τη φάρμα των τρόλ, πώς τους κατασκευάζουν εκεί μέσα από το Κρεμλίνο. Και δεν προσπαθούν να περάσουν όλες αυτές τις διαδικασίες και τα στρώματα της γραφειοκρατίας για να φτάσουν εκεί που χρειάζεται. Ξέρουν το δρόμο. Και είναι και αποτελεσματικοί και ευέλικτοι. Αυτή η ιδέα των τρόλ από την αρχή δεν ήταν να προσπαθήσουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση, αλλά να ε, ρυπάνουν το κυβερνοχώρο. Ε, ξεκίνησε αυτό από το 2005 στη Ρωσία, όταν οι περισσότεροι φιλελεύθεροι ε, δημοσιογράφοι είχαν αποπεμφθεί από τα μίντια και ε, ο μόνος χώρος που μπορούσαν να εκφραστούν ήταν το διαδίκτυο στο παρελθόν είχαμε δελτία ειδήσεων. Μετά έγιναν αυτά blog και πολύ σημαντικά και πολύ ισχυρά. Και τα τρόλ τα, να τα ε, αμολύει το Κρεμλίνο για να τα καταστρέψει αυτά, για να αδειάσει ο κόσμος και να σηκωθεί να φύγει από τις ιστοσελίδες και τα blog. Και σε κάποιες περιπτώσεις το επέτυχαν αυτό πολύ αποτελεσματικά. Μετά το 2014 ε, κατάλαβαν ότι αυτό μπορούν και να το εξάγουν. Και έγιναν και μεγάλα ασφάλματα. Ε, στην Ουκρανία ε, κάπως πέτυχε αυτό, γιατί έχουμε ε, την ίδια γλώσσα, έχουμε ε, κοινέ καταβολές και κοινή ε, παράδοση. Και επιτέθηκαν στη Δύση, ότι ορίστε, η Δύση δεν σας βοηθάει, δεν πρόκειται να γίνεται ποτέ Γαλλία, ούτε καν Πορτογαλία ε, και στην Ανατολική Ευρώπη άρχισαν να υπονομεύουν έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση και, το Ηνωμένο Βασιλείο και τη Γαλλία. Τώρα έχει αυξηθεί αυτό. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή όταν προσπαθούμε να μετρήσουμε και να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των τρόλ. Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται το, το μεγαλύτερο που πέτυχαν ήταν ότι ανάγκασαν όλο τον κόσμο να, συζητήσει, να συζητάει για τη Ρωσία. Το 2016 στη Realpolitik, στην πραγματική πολιτική, πολύ λίγο επέτυχε το Κρεμλίνο και έκτοτε. Παραμένουν οι κυρώσει, οι σχέσει μάλλον Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία δεν είναι καλέ και δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά όλοι για τη Ρωσία συζητάνε. Και ο Πούτιν ανεβάζει, κατεβάζει βασιλιάδες και είναι η χώρα αυτή η πιο ισχυρή στον κόσμο. Υποτίθεται. Στη Ρωσία αυτό δεν είναι μεγάλο ε, θέμα, ούτε εσύ. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό πλαίσιο. Για το περιεχόμενο τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση τι να κάνουμε γι' αυτό. Α είμαστε πρακτικοί. Εγώ σου δημοσιογράφος, ε, πρακτικός άνθρωπος. Έχω δει τόσε προσπάθειες να γίνονται στην Ουκρανία, στη Δυτική Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη. για να αποκρουστεί η online προπαγάνδα και παραπληροφόρηση της Ρωσίας. Και μερικά από τα project αυτά είναι πολύ καλά, αλλά πόσα γνωρίζουμε. Και πόσα χρόνια διαρκούν. Όταν φτιάχνεις ένα αφήγημα και προτείνεις κάτι, ε, σε ένα θέμα και αρχίζει να το συζητάει ο κόσμος. Είναι τελείως διαφορετικό από το να πεις ότι όχι, όχι, ήταν λάθος η είδηση, να σας πω εγώ πώς έγινε, ποια είναι τα προβλήματα. Με αυτό δεν ασχολείται κανένας. Αλλά έχετε δίκιο κυρία Γκόμες, απολύτως. Είναι πολύ ισχυρό το αφήγημα και όλοι θέλουν να το ακολουθήσουν και να... Panama Papers, Paradise Papers, όλα αυτά της ερευνητικής δημοσιογραφία. ανάγκασαν τον κόσμο να συζητάει για τη Ρωσία, για τη διαφθορά, ε, για τα πραγματικά δεδομένα και όντως και στη Ρωσία έγινε κάποιος άλλος. Και αν ρωτήσετε στη Μόσχα τι, τι επίπτωση είχαν τα Panama Papers, άρχισε να αντιδρά ο Πούτιν με μεγάλη προπαγάνδα το 2016 προς τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί αισθάνθηκε ότι του επιτέθηκαν και μάλιστα το επιτελείο της Χίλαρη Κλίντον. Ε, Βεβαίω είναι τεράστιος αντίκτυπος και ως ε, δημοσιογράφος και ρεπόρτερ θεωρώ ότι είναι καλό αυτό γιατί όταν γίνονται έρευνες από πραγματικούς δημοσιογράφους, έγκριτους και αξιόπιστους και όταν αυτά δημοσιεύονται σε βαστά έντυπα και σοβαρές εφημερίδες, τότε μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη ας πούμε σε κάποιους, γιατί βγαίνουν ονόματα επιτέλους και εκεί ε, αυτό δημιουργεί ειδήσει. Πολύ σημαντικό. Για να επανέλθω τώρα στην ερώτηση του κ. Κέλαμ για τη στρατηγική. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, αλλά αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε για τη Ρωσία είναι το εξής. Το Κρεμλίνο όλα αυτά τα χρόνια έτρεμε το διαδίκτυο. Πώς να το πω τώρα. Γιατί όλη αυτή τη στρατηγική, σε αυτό το παιχνίδι όταν μιλάμε για το ίντερνετ και όλες τις νέες τεχνολογίες, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε στρατηγική είχε χαράξει η Σοβιετική Ένωση προ διαδικτύου. Και αυτές οι νέες τεχνολογίες, επειδή κυρίως αναπτύσσονται στη Δύση, ευνηδιάζουν τα δικτατορικά καθεστώτα συνήθως και ψάχνουν πώς θα αντιδράσουν. Και μετά έρχεται το Messenger, μετά έρχεται το VPN. Ε, όλοι τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις, ε, τα δικτατορικά καθεστώτα και φοβάται πάρα πολύ το Κρεμλίνο. Πρόπερση ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε ε, μια νέα στρατηγική για την πληροφόρηση και είναι πάρα πολύ σοβιετική σκοπή αυτό. Και αυτό είναι περίεργο. Πριν έρθουν νέε τεχνολογίε στι τηλεπικοινωνίε στη Ρωσία, οι εταιρείε πρέπει να πάνε πρώτα στι υπηρεσίε ασφαλεία και να ζητήσουν την άδεια. Τι θα κάνουν αυτέ οι νέε τεχνολογίε. Σοβιετικού τύπου πράγματα είναι αυτά. Η εθνική ασφάλεια και οποιαδήποτε ασφάλεια είναι πιο σημαντική από την ανάπτυξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Άρα είναι αδίέξοδο. Και γι' αυτό κατέρευσε ακριβώς η Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τέλος. Υπάρχει όμως μια στρατηγική που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όχι πάρα πολύ καλά ανεπτυγμένη, αλλά βασίζεται σε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Ο Πούτιν είναι πάρα πολύ δημοφιλής στη Ρωσία. Όχι επειδή είναι τόσο τυχερός ή για λόγους οικονομικούς, αλλά από τη δεκαετία του 90 και αρχή του 2000 είδαμε να καταστρέφεται τελείως η εμπιστοσύνη στους θεσμούς στα μάτια των Ρώσων πολιτών. Και το Κρεμλίνο με μαεστρία αυτό το εκμεταλλεύτηκε. Στη Ρωσία κανείς δεν πιστεύει ούτε στα συνδικάτα, ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στους πολιτικούς. Το μήνυμα του, Πολύνου, κάθε φορά, του Κρεμλίνου ήταν να λένε κάθε φορά ότι όλοι αυτοί είναι διεφθαρμένοι και βγήκαν στην πολιτική γιατί θέλουν να πλουτίσουν. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, ότι αφήστε αυτά τα κυβερνητηλίκια στους επαγγελματίες να τα κάνουν και μην τα κάνουν οι πολιτικοί. Και θέλουν τώρα να εξαγάγουν αυτή την ιδέα της έλλειψης εμπιστοσύνη, τη καχυποψία στους θεσμού και προ τη Δύση. Δυστυχώ, αυτό έχει εδώ βάση, γιατί πολλοί κόσμος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που λειτουργούν οι κυβερνήσει και οι διοικήσει στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ. Αυτή είναι η βασική ιδέα, αλλά θα πρέπει να την εντοπίσουμε αυτή την απειλή, να την αγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι τεχνολογίε που χρησιμοποιούν τα τρόλ. Δεν, δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Okay. Colleagues. Συνάδελφοι, έτσι κλείνουμε το σημείο αυτό στη μέση διάταξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τους ευχαριστώ που συμμετείχαν στη συζήτηση. Χειροκρότησε τους παρακαλώ.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 Ναι. Ναι. Colleagues, Καθίστε παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Next point Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι ένα για την αντιμετώπιση των υπηρετικών απειλών. Με χαρά καλωσορίζω δύο εκπροσώπους του Παριζιάνικου Ινστιτούτου, ε, Ινστιτούτο για την Στατικική Έρευνα. Το ξέρουμε εμείς αυτό το Ινστιτούτο. Το εκπροσωπεί ο κύριος Jean-Jacques ανώτατος ερευνητής στο Ίδρυμα αυτό στο Παρίσι και ο δόκτωρ Νίκολας Ματζουκή, ερευνητής στο ίδρυμα αυτό στο Παρίσι. Ο, ο κ. Ματζούκη όμως είναι και εμπειρογνώμονας στα, στην ανάλυση ε, ιδίων θεμάτων για το γαλλικό στρατό. Κύριε Πατχή, έχετε πρώτο το λόγο. Okay, uh, Microphone? ακούτε? Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που σας συναντώ και που θα σας μιλήσω για κάποιες σκέψεις που κάνω για ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Υβριδικές απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων. Τις απόψεις θα ακούσετε να τις θεωρήσετε προσωπικές. Mm. Αυστηρά προσωπικές. Δεν είναι γαλλική επίσημη θέση αυτή που θα σας εκφράσω εδώ. Θα σας κάνω μια ομιλία πάνω σε τέσσερα σημεία. Τι είναι αυτή ο υβριδικός χαρακτήρας του πολέμου, η προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υβριδικές απειλές, η εφαρμογή του στην περίπτωση των ε, Δυτικών Βαλκανίων και κάποια τελικά συμπεράσματα. Το πρώτο σημείο. Για την υβριδικότητα. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Προέρχεται από το στατιωτικό τομέα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δυτικές χώρες ασκούν τον πόλεμο σήμερα και στα τέλη του 20ου αιώνα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι το σημερινό μας θέμα, αλλά εάν δεν μοιράζεσαι αυτές τις δυνατότητες και αν είσαι σε αντίθετο στις δυτικές χώρες, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημά σου είναι πώς θα αντιμετωπίσεις έναν ισχυρό αντίπαλο χωρίς να εκτεθείς θανάσιμα. Αυτή είναι η ιδέα της υβριδικότητας προέρχεται από την ε, επώδυνη εμπειρία των Αμερικανών στο Ιράκ και ε, την Ισραηλινή εμπειρία στο Λίβανο. Πέντε χρόνια χρειάστηκαν για να καταλάβουμε είναι αυτός ο υβριδικός χαρακτήρας του πολέμου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί. Το σίγουρο είναι ότι από γραφειοκρατική σκοπιά το δόγμα αυτό υιοθετήθηκε από τη ΣΥΠΑ το 2010 στην ε, τετραετή αμυντική επισκόπηση. Ε, μετά την Ουκρανική κρίση, η έννοια αυτή, το δόγμα αυτό υιοθετήθηκε από το ΝΑΤΟ το 2015 και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Είναι περίπλοκο γιατί ο Βρετικός πόλεμος σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και στην πραγματικότητα ο συνδυασμός όλων αυτών των ιδεών δημιουργεί τον περίπλοκο χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα μια λέξη μόδας αυτό το hybridity, η υβριδικότητα, ε, για κάτι που υπάρχει πολύ στο διεθνή χώρο, ε, που είναι ε, η επιστροφή του πλήρους πολέμου στις διεθνείς σχέσεις. Σε πολιτικό επίπεδο είναι ε, όταν ε, μία κρατική ή μη κρατική οντότητα αμφισβητεί την ε, διεθνή τάξη δια της βίας με τη δύναμη. Σε στρατηγικό επίπεδο είναι ο συνδυασμός στρατηγικών άμεσων και έμεσων που συμπεριλαμβάνει όλα τα μέσα, συμβατικά και μη συμβατικά και σε τακτικό επίπεδο είναι κάποιες δράσεις συμβατικές και μη συμβατικές, τρομοκρατία κτλ. Ο στόχος της ε, υβριδικότητας να δημιουργήσει μια διαρκή ασυμμετρία στους τρόπους και στα μέσα όταν ε, ας πούμε έχεις απέναντί σου έναν αντίπαλο σαν τη Δύση, μια δυτική χώρα κτλ. Το, θε, το θέμα τώρα είναι γιατί είναι σημαντική η υβριδικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, φυσικά είναι σημαντική για το ΝΑΤΟ. Αλλά δεν μιλάμε για το ΝΑΤΟ σήμερα. Υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση του 2015 για να μελετηθεί το πρόβλημα. Μετά την Ουκρανική κρίση, πολλές χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη, θεώρησαν ότι αντιμετωπίζουν ένα είδος πολέμου. Ε, και ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουν τον πόλεμο αυτό δεν ε, ήταν ε, έτοιμος, δεν ήταν, δεν ήταν αρκετά προετοιμασμένες οι χώρες αυτές. Χρειάζεται μια νέα ανάλυση, μια νέα πραγματογνωμοσύνη, η οποία αναπτύσσεται σιγά σιγά, ε, συμπεριλαμβάνοντας αυτήν την έννοια της υβριδικότητας. Ε, η υβριδική απειλή, υπάρχει ορισμός για αυτήν. Ε, ποια είναι η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες ε, ερμηνείες. Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από αυτόν τον ορισμό της υβριδικότητας. Καταρχάς και πολύ σημαντικό, η υβριδική απειλή αφορά καταρχάς το κράτος, τους κρατικούς φορείς. Δεύτερον, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις τι υβριδικές απειλές σου, Επομένως, μια συντονισμένη απόκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προϋπόθεση. Και τέλος, η κοινή ανακοίνωση έκανε μια πρόταση με 22 δράσεις για να μελετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες της πτυχές του υβριδικού χαρακτήρα του πολέμου. Η υβριδικότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει τώρα στις ευρωπαϊκές, εμπεριέχεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές, υπάρχει ένα κείμενο ε, από το στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το εγχειρίδιο μιλάει για τις διαδικασίες, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δομών που αντιμετωπίζουν ειδικά την υβριδικότητα ε, με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το συμπέρασμα είναι ότι η βρυδικότητα επιβεβαιώνεται ως μείζον πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βραβικό πλαίσιο που προτείνεται το 2016 ε, αναπτύσσεται για να βοηθήσει τις κυβερ... τους κρατικούς φορείς για να εντοπίσουν ποια είναι τα ευάλωτα, ευάλωτοι του, τους, να βρεθούν τεχνικές λύσεις και να συντονιστούν οι απαντήσεις ε, στα πλαίσια ενός σφαιρικού συνολικού όλου. Να αυξηθεί η αντοχή και ανθεκτικότητα των κοινωνιών, όχι μόνο των κρατικών φορέων, των κοινωνιών γενικά και σε στενή συνεργασία να, με, τον, με άλλους εταίρους να γίνουν όλα αυτά και πάνω απ' όλα με τον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων, τι χαρακτήρα παίρνει αυτός ο υβριδικός πόλεμος. Μας μπερδεύει αρκετά. Είναι περίπλοκο, γιατί υπάρχουν πολλά είδη προβλημάτων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν υβριδικά. Το πρώτο είναι πραγματικές απειλές στην εδαφική ακαιρεότητα. Υπάρχει πρόβλημα στα εδαφική ακαιρεότητας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, διεκδικήσεις συνόρων, ε, διεκδικήσεις περιοχών, αλυτρωτικές ε, διεκδικήσεις. Επίσης, ε, πολιτικοί αγώνες για δικαιώματα ε, μειονοτήτων, δημιουργία έντασης λόγω πιθανής απόσχησης ενός τμήματος του εδάφους ή ε, πολιτικά προβλήματα υψηλού διαμετρήματος, ας πούμε. Το δεύτερο είναι μια σειρά κινδύνων, όχι απειλών, το δεύτερο είδος προβλέμου. Πολιτικές, διακρατικές έτσι, προσπάθειες που γίνονται και τώρα επηρεάζονται ε, λόγω του ότι μπλέκονται ξένες, μη ευρωπαϊκές χώρες στην περιοχή. Η Ρουσία, η Τουρκία φυσικά, Σαουδική Αραβία κτλ. Αυτό δημιουργεί μια τελείως διαφορετική έτσι και ανταγωνιστική εικόνα για το μέλλον της, των χωρών αυτών, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης έχουμε και προκλήσεις στις κοινωνίες των χωρών αυτών. Ε, η δημοκρατική διαδικασία, διαδικασία εκδημοκρατισμού, οικονομική ανάπτυξη, μετανάστευση δύο ειδών, Καταρχάς, οι κάτοικοι των Βαλκανίων που πηγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετανάστες από την Μέση Ανατολή. Ε, περνάνε μέσα από τα Δυτικά Βαλκάνια για να φτάσουν στι υπόλοιπε χώρες τη Ευρώπη και τέλος ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Αν πάρεις όλες αυτές τις απειλές, κινδύνου και προκλήσει μαζί, πιθανότατα να μπορεί να πει ότι οι βρυδικέ απειλέ θα μπορούσαν να υποσκάψουν τη διαδικασία διεύρυνση την οποία έχει ξεκινήσει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεσμεύεται απέναντι στις χώρες αυτές. Ας μιλήσουμε τώρα για την στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμόσουμε απέναντι στην υβριδικότητα. Με βάση τόσα υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια διτή στρατηγική σε ιδεολογικό χώρο. Καταρχάς, άμεσο αποκύημα των κριτηρίων Κοπενχάγη Plus είναι ότι αν χρησιμοποιήσουμε το, τις υβριδικές απειλές και τις εφαρμόσουμε στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων και αν θεωρήσουμε ότι η αθεκτικότητα είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές, υπάρχουν δύο τρόποι από τους μπορούμε να επιλέξουμε. Καταρχάς, αθεκτικότητα που σημαίνει να προωθήσουμε αξίες ε, έτσι, ανοιχτών ε, κοινωνιών στις χώρες αυτές των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, στρατιωτικό δυναμικού εδώ και δυνατοτήτων, αλλά εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της μάζας, των μαζών. Και το να προωθήσουμε ιδέες και αξίες μέσω όλων των μέσων που έχουμε. Δηλαδή, μιλάμε για τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τις προωθήσουμε στις χώρες αυτές. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δώσουμε βοήθεια, αρρωγή, τεχνικής φύσεως, στις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν κριτικέ απειλές. Να εντοπίσουμε που είναι, σε ποια σημεία είναι βάλλοντες. Υπάρχουν μέθοδοι και εργαλεία για να εντοπίσουμε τα προβληματικά σημεία και να τα αντιμετωπίσουμε και φυσικά να τους δώσουμε και τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κύριε και κύριοι. Σας δίνω το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατρί. Θα δώσω τώρα το λόγο στο δόκτωρα Νικολά Ματσούκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας παρουσιάσω ε, ε αυτά που έγραψε η δόκτωρη Ζαμπέλ Φακονσιό και μπορεί να το έχετε λάβει. Η παρουσία και η ε, ε, η επιρροή της Ρωσίας στα Δυτικά Βαλκάνια και κάποια άλλα ε, στοιχεία που έχω μελετήσει εγώ για την ενέργεια και το κυβερνοχώρο. Για... τα Ανατολικά Βαλκάνια μιλάει ο μιλητής. Ε, υπάρχει μια επιρροή της Ρωσίας και κάποιοι εθνικιστές εμπειρογνώμονες Ρώσοι λυπούνται για το γεγονός ότι η Ρωσία χάνει τελικά τα Βαλκάνια και ότι η Μόσχα εγκαταλείπει την πρωτοβουλία και χάνει το πάνω χέρι σε αυτή την περιοχή. Αν δούμε κιόλα ε, το τελευταίο δόγμα εξωτερικής πολιτικής ε, της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον Νοέμβρη του 2016, μας αφήνει την εντύπωση ότι τα ανατολικά, δηλαδή δυτικά Βαλκάνια δεν είναι πια προτεραιότητα για τη Ρωσία σε αντίθεση με άλλες περιοχές του κόσμου όπως είναι η Αμερική. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει την πρόθεση να συνεισφέρει καθόλου στην προώθηση της σταθερότητας και την επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή αυτή. Τώρα, αν δούμε ε, πώς τα, βλέπουν αυτά δυτικές χώρες, είναι τελείως διαφορετική αντίληψη, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παρατηρητές που θεωρούν ότι η Ρωσία ενδεχομένω να προετοιμάζεται να υποδαβλήσει κάποιες αιστείες ανάφλεξης και σύγκρουσης για να αποσταθεροποιήσει ε, ή να εμποδίσει με διάφορα μέσα ε, τα δυτικά συμφέροντα να εγκατασταθούν και να ασκούνται στην περιοχή αυτή. Ενισχύες για την ε, θέση της Ρωσίας στη Βαλκανική έχουν ενισχυθεί από μια απόπειρα ε, ε, πραξικοπήματος στο Μαυροβούνιο ε, το φθινόπωρο του 2016 από φιλορώσους Σέρβους εθνικιστές που ενδεχομένως να υποστηρίζονται και από ρωσικά όργανα και οντότητες κρατικές. Οπότε οι δυτικοί ηγέτες όλο και περισσότερο ε, ασχολούνται με αυτή την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και παρακολουθούν πάρα πολύ προσεκτικά τη δράση και τη θέση της Ρωσίας εκεί και ιδιαίτερα στη Σερβία. Όπου, παραδείγματος χάρη, μεταξύ διαφόρων άλλων, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί ως προς την ύπαρξη ενός κέντρου ε, ανθρωπιστικής εκπαίδευσης το 2012 ιδρύθηκε αυτό στην πόλη Νης της Σερβίας που θεωρείται ε, ότι είναι μια αιστεία ε, ρωσικής επιρροής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την επιρροή και την παρουσία της Ρωσίας εκεί. Δεν συμφωνούν, ε, μάλλον δεν υποστηρίζονται πάντα από ε, αποδείξεις συγκεκριμένες. Δεν θα πρέπει να είμαστε ε, συναισθηματικά φορτισμένοι και να το αναλύουμε με πάθος, αλλά να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία της Ρωσίας και τα κίνητρα. Βέβαια, στα κίνητρα της Ρωσίας απορρέουν από μια σχετικά πρόσφατη ιστορία. Σημαντικότερο ήταν το θέμα του κοσυφοπεδίου, διότι η Ρωσία έκανε ό,τι μπορούσε για να περιορίσει ε, την ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου και την ένταξή του στη διεθνή κοινότητα όσο μπορούσε την περιέπλεξε. Είναι αποφασισμένη η Μόσχα να ε, σταθεί αντιμέτωπη όπου μπορεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δείξει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη Δυτική Βαλκανική. Και πάντα από τη σκοπιά της Μόσχας η διεθνής ε, τάξη έχει περάσει σε μια μεταδυτική εποχή, με την επάνωδο δηλαδή της ισχύω της Ρωσίας και αυτό επιτρέπει στη Ρωσία να προβάλλει τη δύναμή της και να παρουσιάζεται ως μια δύναμη που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Ε, τα Δυτικά Βαλκάνια λοιπόν ε, για πολύ καιρό ήταν ε, προνομιούχα περιοχή για την έκφραση της ε, ρωσικής κυριαρχίας. Και υπάρχουν κάποιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια όπου εκφράζεται αυτό και προάγεται η ρωσική κουλτούρα και ο πολιτισμός από, από ομοσπονδιακές οργανώσεις όπως είναι το Ρώσο Τρουνιτσιέσβο και είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ρωσικού και μεταξύ άλλων είναι επιφορτισμένο με την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας για τη Ρωσία στο εξωτερικό. Από το 2011 είναι στην Κροατία, ε, Μαυροβούνιο και Σλοβενία και από το 2016 στη Μακεδονία, λέει ο και ε, το Ρούσκι Μύρ από το 2009 στην ε, περιοχή εκεί και στη Ρεπόμπλικα Σέρψκα του, ε, της Βοσνίας από το 12. Το 2014 το Σπούτνικ που γνωρίζετε όλη τη σημασία του για ε, κάποια μηνύματα που εκπέμπει από τη Ρωσία ε, άρχισε να εκπέμπει ε, σε διεθνές κανάλι στα σερβικά. Υπάρχουν χώρες πολλές λοιπόν δυτικών Βαλκανίων, Βοσνία, Ζεγοβένη κυρίως και Σερβία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ε, στάση σχετικά θετική και φιλική σε σχέση με τη Ρωσία. Ιδιαίτερα στη Σερβία. Είναι πολλοί εκείνοι που εκφράζουν ικανοποίηση από το γεγονός ότι βλέπουν τη Ρωσία να έχει μια διεθνή παρουσία και στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό που θεωρεί η Σερβία ε, ότι έχει υποστεί αδικία όταν κατέρευσε η πρώην Ιουγκοσλαβία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Ρωσία ότι δημιούργησε ε, αυτή την κόπωση ε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις συγκεκριμένες χώρες. Αλλά είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι το εκμεταλλεύτηκε αυτό μερικές φορές. Άρα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μερικά γεγονότα και να αξιολογήσουμε, να διασταυρώσουμε το αληθοφανές τους, το αληθές τους αυτό το περίφημο ανθρωπιστικό κέντρο της ΝΙΣ θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση παραστρατιωτικών ομάδων και τη σύστασή τους ε, που ήταν ε, πιστά στο Ντόντιτς, ο οποίος ε, ήταν ο εμπνευστή του πραξικοπήματος στο Μαυροβούνιο με την υποστήριξη υποτιθέμενη της Ρωσίας. Επίσης, θα πρέπει να αναλύσουμε και την επιρροή που δεν έχει η Ρωσία στην ενέργεια. Πολύ συχνά προβάλλεται ως προνομιούχος τομέας ρωσικής επιρροής. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε ότι η Ρωσία ουσιαστικά όλο και περισσότερο ε, αντισταθμίζεται εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια, στα ενεργειακά, από άλλες εξωευρωπαϊκές δυνάμεις, και υπάρχει και προμήθεια που μπορεί να έρχεται από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον ίδιο τρόπο το εξωτερικό εμπόριο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με τη Ρωσία τελικά είναι σχετικά περιορισμένο, διότι ε, ανέρχεται στο 6,6% μόλις των Δυτικών Βαλκανίων και 1% του ρωσικού εμπορίου. Βεβαίως ε, η Σερβία είναι ο πρώτος εταίρος και προβάλλεται ως τέτοιος πρώτος οικονομικός εταίρος της Ρωσίας στην περιφέρεια εκεί. Κατά τον ίδιο τρόπο η Ρωσία τελικά είναι επενδυτής σχετικά μικρός. Γιατί σε ό,τι αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις της Ρωσίας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Ακόμα και στη Σερβία το μερίδιο της Ρωσίας στις ξένες άμεσες επενδύσεις ε, ανέρχεται μόλις το 4,9 και 3,6% ετησίως σε σχέση με το 70-80% που είναι το οι επενδύσεις μάλλον από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν έχει ισχυρή επενδυτική παρουσία τελικά η Ρωσία. Και η οικονομική παρουσία της Ρωσίας που μπορεί να φαίνεται σχετικά υψηλή δεν απέτρεψε κάποια πράγματα. Ας πούμε στο Μαυροβούνιο έχει σημασία να τονίσουμε ότι το 1 τρίτο των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στο Μαυροβούνιο συνδέονται με τη Ρωσία. 25% των τουριστών είναι Ρώσοι και 7.000 Ρώσοι διαμένουν μόνιμα στο Μαυροβούνιο. Αυτό δεν ε, εμπόδισε το Μαυροβούνιο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα. Ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τη γλώσσα επίσης που συχνά χρησιμοποιείται ως φορέας ε, επιρροής η, Ρωσία δεν έχει και τόσο τεράστια ε, επιρροή ή πλεονέκτημα γιατί η ρωσική γλώσσα δεν ομιλείται τόσο πολύ στην περιοχή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πιστεύουμε συνολική στρατηγική της Ρωσίας στη συγκεκριμένη περιφέρεια αλλά ευκαιριακό τρόπο δρά ή σχετικά ευκαιριακό κάθε φορά. Και η αρχή για τη Μόσχα ε, είναι να χαλάει λίγο ε, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Μόσχα έχει επίγνωση του ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική για τις χώρες αυτές από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δραστηριοποιείται πραγματικά στο δυσκολεύει τη διεύρυνση και να την κάνει όσο γίνεται πιο περίπλοκη. Και τέλος, euh, ε, και έχει ένα οπορτονιστικό ρόλο ε, αποσπασματικό και συγκεκριμένο. Να σας εξηγήσω λοιπόν όλα αυτά, τα οποία δεν ήταν δικά μου, αλλά ήταν της δόκτωρος που είχε ετοιμάσει το έγγραφο για τη Ρωσία, θέλω να επιμείνω σε μερικά σημεία που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά, που συχνά προβάλλονται ως κεντρική ιδέα για την εξάρτηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων από τη Ρωσία. Αν δούμε εδώ τις εισαγωγές από τη Ρωσία των κρατών αυτών, τι διαπιστώνουμε. Με εξαίρεση τη Σερβία, τη Σλοβενία και τη Βοσνία, Ριζεγοβίνη, όλες οι υπόλοιπες χώρες εμφανίζουν σταθερή ε, εξάρτηση από εισαγωγές ή μείωση. Και όλο και περισσότερο μπαίνουν άλλοι παράγοντες ε, και ε, στο, στα πετρελαϊκά και στα θέματα του φυσικού αερίου και των αγωγών στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό ε, υποστηρίχθηκε και από μια επιθυμία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εξοκοινοτικών παραγόντων, κυρίως το Ζερμπαϊτζάν που δίνει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και η Τουρκία που είναι διαμεσολαβητής και περνάνε η αγωγή φυσικού αερίου και έρχονται και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο αυτοί για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αν κοιτάξετε εδώ πώς έχουν σήμερα η αγωγή και τα μελλοντικά έργα για ε, το φυσικό αέριο, διαπιστώνουμε ότι η σημερινή διάρθρωση αγωγών φυσικού αερίου ε, εξαρτάται πάρα πολύ από τη Ρωσία σήμερα, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τις διασυνδέσεις των αγωγών φυσικών αερίων, του αγωγού Transbalkan που περνάει από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ή το κεντροευρωπαϊκό δίκτυο που περνάει από την Ουκρανία και καταλήγει στην Αυστρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τον νότιο διάδρομο ακριβώς θέλει να ευνοήσει και να προωθήσει εναλλακτικό δρόμο ε, προμήθειας που περνάει τώρα από την Τουρκία για το αέριο από το Αζερβαϊτζάν με ένα διπλό σύστημα ΤΑΝΑΠ λέγεται ο αγωγό στην Τουρκία και ΤΑΠ ε, ε, από την Ελλάδα, την Αλβανία και καταλήγει στην Ιταλία και περνάει την Αδριατική. Αυτός ο αγωγό ΤΑΠ λοιπόν είναι ένα νέο έργο και είναι ένας αγωγός που περνάει από τα Βαλκάνια, μετά στην Ιταλία και φτάνει μέχρι την Κροατία. Με αυτό το νέο διάδρομο λοιπόν για το φυσικό αέριο ευνοούνται νέοι παράγοντες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον απλούστατο λόγο ότι ο ΤΑΠ, ο αγωγός αυτός που φέρνει από το Αζερβαϊτζάν το φυσικό αέριο μέσω της Τουρκίας και σε μεγάλο βαθμό είναι η δοξησία Σοκάρ που είναι η αζέρικη εταιρεία αλλά και εξαρτάται και από την καλή βούληση της ε, Τουρκίας και υπάρχει και ο αγωγός ΙΑΠ που είναι Ιωνίου και Αδριατικής. Ε, αυτά ε, είναι όμιλοι κυρίως των Δυτικών Βαλκανίων σε συνεργασία με τη ΣΟΚΑΡ, την Αζέρικη εταιρεία. Άρα μειώνεται η επιρροή της Ρωσίας και έρχεται να αντισταθμιστεί από την επιρροή άλλων παραγόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής γενομένης εδώ από το Αζερβαϊτζάν, αλλά και την Τουρκία, η οποία όλο και περισσότερο ανεβαίνει και είναι παρούσα και ως προς τη βιομηχανία και ως προς την ενέργεια σε κάποιες χώρες, Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο. Αντίστοιχα, εάν δούμε τι γίνεται τελικά με την επιρροή στον κυβερνοχώρο, τι διαπιστώνουμε, ότι η θέση της Ρωσίας γενικά στα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι και τόσο σημαντική, διότι αν κοιτάξουμε την επιρροή και την παρουσία ε, ρωσικών ιστοσελίδων ε, στα Βαλκάνια και στο κοινό, βασικά στο Μαυροβούνιο είναι ε, μεγάλη. Και η πρώτη ιστοσελίδα που κοιτάνε είναι το F-Contact είναι περίπου το ρώσικο Facebook, αλλά είναι το, η ενδέκατη πιο δημοφιλής σελίδα στο Μαυροβόνιο και εκεί θα πρέπει να σχετικοποιήσουμε λίγο την επιρροή τους και πόσο η Ρωσία δρά στο διαδίκτυο. Γιατί χώρες αυτές, έξι χώρες, έχουν ένα ντόπιο οικοσύστημα στον κυβερνοχώρο και στο διαδίκτυο και έχουν αυξήσει και τις δυνατότητές τους, έτσι ώστε να μπορούν να θεωρούνται ορισμένες από τις χώρες αυτές ε, πολύ ανθεκτικές, παράδειγμα, για τον κυβερνοχώρο πάντα. Υπάρχει ένας διεθνής δείκτης του Διεθνούς Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών και η Κροατία είναι στη θέση 41, που είναι πάρα πολύ καλή ε, ως προς την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Άρα λοιπόν είναι περιορισμένες οι δυνατότητες και της Ρωσίας αλλά και η περιοχή και κάποιων άλλων παραγόντων. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ. Συζήτηση τώρα. Ο κύριος Νταζάν πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας που βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες και με στοιχεία. Δεν έχω τόσο ερωτήσεις όσο παρατηρήσεις. Εμπεριστατωμένες ήταν οι μελέτες Όσον αφορά τον ευρυδικό χαρακτήρα, καλά το συνοψίσατε τη συζήτηση. Ε, πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτός ο όρος γιατί είναι το αλατοπίπερο, πάει σε, στα πάντα. Ε, από πλευράς marketing, ε, όντως έχει μεγάλη επιτυχία. Ένα σωρό συνέδρια γίνονται με αυτό το θέμα και δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό τομέα, αφορά και το μη στρατιωτικό. Ε, πάντως έχετε δίκαιο που λέτε ότι είναι μια νέα ορολογία για ένα φαινόμενο όμως που δεν είναι νέο. Υπάρχει η στρατηγική πτυχή, η τακτική πτυχή. Αυτά δεν είναι καινούρια και καλά κάνατε και πήρατε για παράδειγμα τα Βαλκάνια σήμερα. Όμω, ο πόλεμος στα Βαλκάνια, τέο Γιουγκοσλαβία, τι έκανε ο Μιλόσεβιτ στη δεκαετία του 80 και του 90, είναι ακριβώς αυτό το υβριδικό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε για τον κυβερνοχώρο, αλλά η προπαγάνδα, οι πόλεμοι μέσω εξουσδότηση, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα είχαμε ήδη. Άρα τον ευρυδικό χαρακτήρα τον βρίσκουμε ήδη στη Γιουγκοσλαβία της δεκαετίας του 80 και του 90. Και από εκεί και πέρα όλες οι άλλες οι ιδέες που προστίθονται ε, μας φαίνονται κάπως αστείες. Τώρα για τη σημερινή κατάσταση. Η ανάλυση της κυρίας Φαλκό παρά είναι ορθολογική. Ενώ ακριβώς μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βασίζεται περισσότερο στη ρητορική, στην αντίληψη, στην προπαγάνδα, στην επιρροή και όχι τόσο σε ε, δεδομένα, σε γεγονότα. Ενέργεια, για παράδειγμα. Έχετε δίκιο ενεργειακές ε, ροές. Δεν είναι τόσο πολύ υπέρ της Ρωσίας. Εν μέρη έχει σημασία αυτό. Αλλά να δείτε στη Σερβία. Την επιχείρηση της ΝΙΣ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις υπηρεσιών. Ο οικονομικός μοχλός, ο κοινωνικός μοχλός από αυτή την επιχείρηση είναι τεράστιος. Πώς Σέρβοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, οι ίδιοι μέσω των οικογενειών του συνδέονται με την ΝΙΣ, με τα ταμεία της. Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο μοχλό. Πολύ περισσότερο από τους τόνους πετρελαίου που εισάγεται. Όταν λέτε ότι υπάρχουν διακλαδώσεις σήμερα που μας οδηγούν αυτονομούμεθα απέναντι στη Ρωσία, ναι και όχι. Γιατί άλλες επιχειρήσεις άλλων τρίτων χωρών επίσης έχουν ρωσική επιρροή. Οι Ούγγροι μέσω της Μόλ για παράδειγμα, οι άλλοι χώρες δηλαδή που εκ πρώτης όψης φαίνεται να μην εξαρτώνται από την Ρωσία, Κροατία για παράδειγμα, και όμως η Κροατία έχει τεράστια ρωσική επιρροή και ανησυχούν οι ίδιοι οι Κροάτες πολιτικοί. Γιατί τη βλέπουν, βλέπουν τους ολιγάρχες, βλέπουν τους ενδιάμεσους και όταν το ψάξουμε διαπιστώνουμε ότι λίγο πολύ η επιρροή είναι από τη Ρωσία. Υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα, υπάρχουν ε, τα στατιστικά, αλλά υπάρχει και ολόκληρη αυτή η επιρροή που έρχεται πιο διακριτικά, που διαχέεται αλλά που είναι σημαντική. Εξού και αυτό που λέτε για τα μέσα ενημέρωσης, κυβερνοχώρος, διαδίκτυο κλπ. Στο Μαυροβούνιο, εντάξει, μα δεν χρειάζεται να πάει κανείς σε ρώσικες ιστοσελίδες, έτσι κι τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα αυτή είναι ρωσικής επιρροής. Και συνεχίζουν δομές που υπήρχαν πριν και που χρηματοδοτούνταν από τη Ρωσία. Στα Βαλκάνια το βασικό είναι ότι οι χώρες αυτές έχουν μνήμη που εμείς δεν έχουμε. Στις χώρες αυτές έχετε δίκτυα τα οποία δεν διαλύθηκαν ποτέ. Διάφοροι συνάδελφοι λένε «Μα δεν υπάρχει απόδειξη στα βακάνια, δεν φαίνεται αυτό». Ναι, μα έχετε μια χώρα η οποία διαλύθηκε, αλλά αυτά τα δίκτυα τα σκοτεινά, γιατί υπήρχαν έτσι στη Γιουγκοσλαβία, αυτά τα δίκτυα λοιπόν δεν διαλύθηκαν ποτέ. Παραμένουν λίγο ή πολύ. Εμείς δεν τα θυμόμαστε αυτά. Οι δυτικοί, οι αξιωματούχοι, οι Ευρωπαίοι που πάνε και διαπραγματεύονται με τη Βοσνία, το Κοσμοπέδιο κτλ. Ε, άντε, το 99 λιγάκι να ξεκίνησαν με τον Άτο, νωρίτερα κανένας δεν είχε ασχοληθεί με Κωσυφοπέδιο και τέτοια. Οι ηγέτες όμως της περιοχής την έχουν αυτή τη μνήμη και εδώ και 30 χρόνια μας βλέπουν να δείχνουμε ενδιαφέρον για αυτούς. Αυτοί όμως εξακολουθούν να έχουν τα συμφέροντά τους που παραμένουν τα ίδια και που δεν είναι απαραίτητα συμβατά με τα δικά μας. Όταν λοιπόν σήμερα λέμε ότι θα πάμε και θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, θα πάμε να τους μάθουμε πράγματα, ε, νομίζω ότι εδώ δεν μετράμε καλά τα πράγματα. Για αυτούς το θέμα της αντοχής δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό και εγώ είμαι πιο εντάξει, προβληματισμένο, δεν θα έλεγα πεσιόδοξος, αλλά πιο προβληματισμένο. Και όταν λέμε ότι η Ρωσία δεν έχει στρατηγική και οπορτουνιστικά άδρα, το λέμε αυτό πολύ εύκολα για όλου και για τα Βαλκάνια κλπ. Όχι, μπορεί να μην έχει στρατηγική η Ρωσία, αλλά προχωράει σε όλα τα μέτωπα. Και μαζικά και καλά συντονισμένα, από ό,τι φαίνεται όσον αφορά τον κρατικό μηχανισμό. Οπότε είναι αυτό ο οπορτουνισμός, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση για να καλύψουμε τη δικιά μας έλλειψη στρατηγικής, γιατί από πλευράς δικιάς μας, θετικών χωρών, τι διαπιστώνουμε. Δεν αλλάζουμε εμείς το παιχνίδι. Η ικανότητα ε, να δημιουργήσει αλλαγές η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σήμερον ημέρα δεν υπάρχει πια. Ε, η Κομισιόν προσπαθεί, εντάξει, δημοσιεύει στρατηγική για τα Βαλκάνια, αλλά δεν υπάρχει πολιτική πνοή, δεν υπάρχει πραγματική στρατηγική. Υπάρχουν κάποια μέτρα, το οποίο εντάξει δεν λέω ότι δεν είναι καλά, αλλά δεν είναι στρατηγική αυτό. Λέμε ότι οι Ρώσοι δεν έχουν, εγώ νομίζω ότι σήμερα έχουν περισσότερο οι Ρώσοι στρατηγική για τα Βαλκάνια από ό,τι έχουμε εμείς. Και οι Τούρκοι μάλιστα, επίσης. Οι Κινέζοι περισσότερο από εμά. Άρα δεν είναι μόνο οι Ρώσοι που παίζουν στα Βαλκάνια. Εμεί τα χάνουμε τα Βαλκάνια, αλλά τα χάνουμε επειδή δεν έχουμε μνήμη, επειδή είμαστε αφελείς, επειδή δεν καταλαβαίνουμε ακριβώ με τι έχουμε να κάνουμε και γιατί προβάλλουμε σε αυτού κάποια μη ορθολογική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. μετά από αυτά που είπε ο κ. Ντονζό, τα οποία ήταν πολύ σωστά διατυπωμένα, θα ήθελα να μιλήσω ξανά για τον ορισμό. Για την ε, ετικέτα που βάζουμε σε μια πολύ παλιά στρατηγική, η οποία ποτέ δεν έχει σταματήσει να υπάρχει, έτσι. Υπάρχουν δίκτυα, ιστορικά δίκτυα, τα ξέρουμε, τα αντιμετωπίζουμε γενικά όπου τυπώνουν διάφορες ανακοινώσεις, ε, έχουν διάφορες στρατηγικές. Ε, μας βοηθάει ίσως αυτή η ετικέτα, γιατί εστιάζει την προσοχή μας και τη δράση μας ίσως. Και συντονίζει λιγάκι στις, ε, συντονίζει λιγάκι ενεργειές μας. Το δεύτερο που θέλω να πω Μετά από αυτά που ο κύριος Πατρί για αυτή την διπτή στρατηγική. Το πρώτο σκέλος αυτής της στρατηγικής είπατε ότι η ανθεκτικότητα σημαίνει πρόθεση αξιών. Μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Ντονζό, θέλω να πω ότι θα πρέπει θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε καλύτερη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει να προωθήσουμε αποτελεσματικά τις αξίες μας. Δεν είμαι σίγουρη το κάνουμε αυτό καλά. Α, δεν νομίζω ότι τα πάμε καλά σε αυτό το μέτωπο. Επίσης, Κύριε Μαζούκη, μιλήσατε για τα θέματα ενέργειας. Και αυτό συνδέεται με κάτι που είχε ο κύριος Πατρί για τους άλλους φορείς. Όλοι αυτοί οι νέοι και καλά φορείς που μας μιλήσατε, ε, που μας είπατε, στην πραγματικότητα είναι παμπάλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κτλ. Το είπε και ο κύριος Ντοζό και αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάντως για τις παρουσιάσεις που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανένας άλλος το λόγο. Άρα, να θέσω κι εγώ μία ερώτηση. προς τον κύριο Ματζούκη. Αλλά ίσως και οι δύο μιλητές θα μπορούσαν να απαντήσουν. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για τη Σερβία. Δεν καταλαβαίνω πλήρως. Το γιατί πρέπει να φέρουμε αυτή τη χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να την εντάξουμε το συντομότερο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για θέματα ασφάλειας και άμυνας υπάρχουν προβληματικά θέματα με την Σερβία. Στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία, κοινά γυμνάσια, κοινέ ασκήσεις στη Λευκορωσία με την Ρωσία. Απ' την άλλη η Σερβία είναι πολύ δραστήρια σε ειρηνευτικές αποστολές στη Δύση, μαζί με τη Δύση. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Έχει συμφωνία πλαίσιο στα, στα πλαίσια της CDA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, Οργανισμό Άμυνας. θα ξεριζώσουμε αυτή τη θέληση που έχει η Σερβία για, να, για συνεργασία με τη Μόσχα σε αυτούς τους τομείς. Μας, εν, μας ενοχλούν αυτές οι επιθετικές πολιτικές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όχι ειδικά για τα Βαλκάνια, αλλά να σας πω την προσωπική μου άποψη η Σερβία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Ρωσία για να αποκτήσει ισχύ απέναντι στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες και να παίξει με στρατηγικές που χρησιμοποιούν και άλλες χώρες στα, Βαλκάνια. Χρησιμεύει ε, ως χώρα διαμετακόμισης για το ρωσικό αέριο προς άλλες χώρες, όπως ας πούμε προς την Βοσνία ζεγοβιν και να εκμεταλλευτεί την ε, σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ρωσία είναι σαν ο μεγάλος αδερφός, ας πούμε, που βοηθάει τη χώρα για να παραμείνει η πιο σημαντική χώρα στην περιοχή. Το πρόβλημα είναι ότι η Σερβία βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίπαλη δύναμη που θα υποσκάψει τη δική της ισχύ στην περιοχή. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιστρέψει αυτό το αφήγημα. Ε, και φοβάται μάλιστα η Ρωσία, η, συγγνώμη, η Σερβία, ότι θα, την, θα υποσκάψει και τη δύναμή της ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αντίθετα η Ρωσία ενισχύει αυτόν τον προσανατολισμό. Είναι, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, ε, είναι ένα αφήγημα ας πούμε της Σερβίας που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιστρέψει, να ανασκευάσει. Γιατί, για το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σερβία. Μάλιστα. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Μπορείτε να κάνετε λοιπόν κάποιε παρατηρήσει ε, με την ίδια σειρά με την οποία πήρατε το λόγο αρχικά. Ο κύριο Πατρί πρώτο. Μικρόφωνο. Deux choses. La première... Να σας πω τα εξής. Καταρχάς, υπάρχει μια παρεξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο μίλησα όταν μίλησα αγγλικά. Αυτό που σας, αυτό παρουσίασε ως τη δυτή στρατηγική είναι αυτό που έχουμε οικοδομήσει με βάση τις διάφορες δομές που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κάποιες δυσκολίες για τη διασύνδεσή τους, ας πούμε, και τη σχέση των διαφορών φορέων. Αλλά αυτό συστήνει, συστήνουν επίσημα τα διάφορα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, το, το, η επίσημη, ας πούμε, συνεργασία. Ε, επίσης, δεύτερον, δεν υπάρχει υβριδική απλή παρά μόνο αν, υπάρχει σύγκρουση, πόλεμος. Για την Ουκρανία, ναι βέβαια. Για τη Συρία και το Ιράκ, ναι. Για την Ιεμένη, ναι. Για τα Βαλκάνια όμως όχι. Δεν υπάρχει πόλεμος στα Βαλκάνια και σήμερα κανένας δεν θέλει να δημιουργήσει νέα ανάφλεξη. Αν λοιπόν τα όπλα είναι ιδεολογικά για να αντιμετωπίσουμε ας πούμε τα διάφορα, τις διάφορες πτυχές της ε, υβριδικότητας στο, στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα, αλλά στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί μπορεί να θεωρήσετε ότι υπάρχει μια γενικευμένη σύγκρουση σε μια περιοχή που υπάρχουν πολλές εντάσεις ήδη. Το να τονίζουμε τις υβριδικές απειλές στα Βαλκάνια, βασικά ε, θρέφει, ας πούμε, της ιδεολειψίας διαφόρων κυβερνήσεων που έχουν αντιπάλους πολύ κοντά στην περιοχή τους, στην περιοχή εκείνη. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μέσω της φύσης τους κτλ, θα έπρεπε να έχουν ως σκοπό όχι να θρέψουν αυτές τις εντάσεις, αλλά να τις μειώσουν. Το να σκεφτούμε ότι, ε, υπάρχουν υβριδικές απειλές, ε, στην πραγματικότητα ε, δημιουργούμε καταστάσεις όπου ε, κάποιοι συντάσσονται με την Ευρώπη, κάποιοι με τη Ρωσία, κάποιοι με την Τουρκία κτλ. Εάν θέλουμε να εστιάσουμε στην υβριδική απειλή πρέπει να έχουμε και θάρρος. Γιατί αυτό που προκύπτει από αυτή τη σύντομη συζήτηση είναι ότι δεν μιλάμε πια για οικονομική ανάπτυξη απλώς. Αυτά τα λέγαμε το 90 και οι αντίπαλοι μας στα Βαλκάνια, από ό,τι ξέρω, είναι, είναι ποιοι. Οι Τούρκοι που δεν είναι τρίτος κόσμος, η Ρωσία που δεν είναι τρίτος κόσμος, η Σαουδική Αραβία ούτε και αυτή είναι τρίτος κόσμος. Αυτά τα μοντέλα κοινωνιών σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη με άλλες αξίες απόλυτα συμβατέ με τις δικές μας. Ασύμβατες. Και Εάν θεωρήσετε ότι θέλετε να κατακτήσετε Βαλκάνια, ας πούμε, τότε θα πρέπει να κάνετε ένα ιδεολογικό πόλεμο ε, τύπου ψυχρού πολέμου. Και εμείς έχουμε αξίες που πρέπει να υπερασπιστούμε στα Βαλκάνια και αν θέλουμε να τις υπερασπιστούμε κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ομιλία μας. Και σας δίνω το λόγο. Έχω, ε, τονίζοντας ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και ως Ματζούκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο για να απαντήσω στα σχόλιά σας ως προς τα ενεργειακά δεν αρνούμε. Μάλλον δεν λέω εγώ ότι σταμάτησε η ρωσική επιρροή στα ενεργειακά, το αντίθετο. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ε, ότι υπάρχει μια μετάβαση του συστήματος. Αρχίσαμε από ένα ενεργειακό σύστημα στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου υπήρχε η Ιουγκοσλαβία, ένα ενιαίο σύστημα μέσω της Σερβίας ερχόταν από τη Ρωσία και ήταν ενιαίο. Τι έχει γίνει όμως τώρα. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, και τη Συμφωνία ε, για την Ενεργειακή Ένωση, τον Νότιο Διάδρομο, δημιουργούνται εναλλακτικέ ε, οδοί ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη των Βαλκανίων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλες πηγές εφοδιασμού. Τώρα είναι το Αζερβαϊτζάν στο νότιο διάδρομο. Αυτό δεν έρχεται να καταργήσει αυτό που προϋπήρχε. Στην υπάρχει η Gazprom Neft, ε, που έχει εργοστάσιο. Ε, και συμφωνώ απολύτως στην ε, οικονομική του αρχιτεκτονική. Ωστόσο, μπορεί να αντισταθμιστεί αυτή η ισχύ εκεί. Με την Ενεργειακή Ένωση τι βλέπουμε. Το σύνολο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έχουν αρχίσει προσπάθειες ή έχουν δηλώσει την πρόθεση να δημιουργήσουν όλο και περισσότερο ένα σύστημα που να βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά γίνονται με ευρωπαϊκές εταιρείες. Αν δούμε ε, στο διαδίκτυο ποιοι είναι οι υπάροχοι των τηλεπικοινωνιών σε όλα τα συστήματα, έχουν ανοίξει με κάποιες εξαιρέσεις και βλέπουμε εκείνοι που δίνουν το διαδίκτυο, οι να είναι Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει πάροχος ε, παροχής διαδικτύου Ρώσος, πολύ σημαντικό στα Δυτικά Βαλκάνια. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα επιρροής εκεί από την, Ευρωπαϊκή, από την Ρωσία. Ε, δεν είναι ένα το σύστημα που ήταν το παρελθόν και κληρονομιά του ψυχρού πολέμου, όπου αναγκαστικά όλα περνούσαν από εκεί. Μπορούν να αντισταθμιστούν και από εναλλακτικέ πηγές. Και όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει εκεί, αλλά και άλλοι φορείς. Αναφερθήκατε στην Τουρκία, αλλά υπάρχει και η Κίνα, το Αζερβαϊτζάν που είχε τεράστια πολιτική επιρροή στα τελευταία χρόνια όταν ήταν πολύ ψηλέ τιμέ του πετρελαίου. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορούν να επηρεάσουν αυτοί οι παράγοντες. Όπως είπαν όμως και οι συνάδελφοι, τελικά τα ευρεδικά ζητήματα είναι ε, η ποιος ασκεί επιρροή και ποιος την αποκρούει. Δεν λέμε ότι υπάρχει το ένα και δεν υπάρχει το άλλο. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Θα υπάρξουν διάβλη σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Έχουμε και εναλλακτική και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη. Σας ευχαριστώ. Very much Εγώ σας ευχαριστώ. Uh, Με την παρατήρηση αυτή ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη που ήταν η ακρόαση για τις uh, υβριδικές απειλές στα Δυτικά Βαλκάνια. Να χειροκροτήσουμε μαζί τους εξαίρετους ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 11 και θα αρχίσουμε στις 9 το πρωί ακριβώς. Κλείνει το μικρόφωνο της Πρόεδρου, δεν ακούμε τι λέει.